Colleagues, good evening. We can give start to the... Συνάδελφοι, καλησπέρα. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Ξεκινάμε σήμερα το απόγευμα και θα μιλήσουμε για τη χρονιά ηθαγένειας το 2013 και επίσης την ε, καμπανία της Ιταλίας, τα απόβλητα με περιφερειακές αρχές και με παρουσία αναφέροντος και επίσης για την αεροκυκλοφορία στην Ισπανία, την μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής της αλληλευτικής πολιτικής ε, με διάφορους φόρους που θα συμμετάσχουν, όπως επίσης και με εκπροσώπους ορισμένων από την Επιτροπή Αλίας και από ορισμένα εθνικά κοινοβούλια και αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε για την έκθεση Βάλιαν. Μετά από τις ανακοινώσεις αυτές, παρακαλώ συνάδελφοι, έχετε μια κάποια παρατήρηση, είτε θεωρούμε ότι εγκρίνεται η μερισιά διάταξη. Καμία αντίρρηση, εγκρίνεται λοιπόν η μερισιά διάταξη. Από πλευρά ε, του συναδέλφου Τσίστερν, Κάσμαν ε, και Μέγερ μου γνωστοποίησαν ότι θα απουσιάσουν ε, γιατί έχουν άλλα καθήκοντα και για τη βάλια θα διεξαχθεί αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο και θα μπορούσε να διεξαχθεί η ψηφοφορία ηλεκτρονικά γι' αυτό παρακαλώ συνάδελφοι να έχετε μαζί σας τις ε, κάρτες σας και εάν έχετε μια κάποια δυσκολία για να ψηφίσετε, μη μάλλον ε, αν θέλετε να την αντικαταστήσετε, να το πείτε στη γραμματεία. Και ακόμα για το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, για τώρα το απόγευμα, θα ήθελα να χαιρετήσω τις αρχές που παρίστανται τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο δόκτωρ Φάλτεμπεργκ, να το χαιρετήσω, και ο Επίτροπος Βοτόσνικ είπε ότι δυστυχώς δυνατή να παραστεί σήμερα το απόγευμα, άρα λοιπόν ο κύριος Φάλτεμπεργκ τον εκπροσωπεί από την περιφέρεια της Καμπανίας στην Άπολη της Ιταλίας έχουμε ακριβώς τον δόκτωρ Ραϊμόντο Σαντακρότσε και από το Δημοτικό Συμβούλιο από κυρία Τσελέστε Τάραντο και επίσης εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής από το Αβελίνο στην περιοχή πάντα, εκεί πάντα το Δημοτικό Σύμβολο Γκαμπακόρτε και το δόκτωρο Πελίτσιο Ντελούκα και από το Σαλέρνο Τζοβάνι Φορτουνάτο και Τζουζέπε Ντακούντσι για το Μπενεβέντο ο Δημοτικός Σύμβολος Τζανλούκα Τσέτο και από την Καζέρτα Μα είχαν ανακοινώσει ότι κάποιος θα ερχόταν, αναφέρεται σημειώθηκαν δυσκολίες, γι' αυτό δεν έχουμε κάποιον από την Καζέρτα. Από την Νάπολη τώρα, κανονικά θα έπρεπε να παρίσταται ο αντιδήμαρχος Σοντάνο, δεν τον βλέπω όμως στην αίθουσα. Μόλις μου είπαν και συγγνώμη για την επαρχία της Νάπολης Τζοβάνα Ναπολιτάνο. Για τους αναφέροντες είναι ο κ. Ματρόνε παρόν που υπέγραψε μια αναφορά επίσης με πάνω από 2.000 ακόμα υπογραφές και σε λίγο θα έρθει και εκείνος για το σημείο 7 τώρα που έχει να κάνει με τους ελεκτές ανέρας κυκλοφορίας στην Ισπανία θα ακούσουμε δύο εκπροσώπους από τους πολλούς που υπέγραψαν την 431 και 651 του 2010, τις αναφορές αυτές. Στις 5.30 θα έχουμε μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών και αύριο το πρωί θα συζητηθούν ε, οι αναφορές ε, για την ε, κοινή ελληνική πολιτική. Για το σημείο 10 για το Παγκόσμιο Ταμείο τη Φύση την 802-2011 αναφορά για την κοινή αλλιευτική πολιτική και ακόμα έχουμε και άλλες αναφορές σχετικά αλλά δεν θα εξεταστούν πάντως ε, είναι παρόμοια το θέμα. Μετά από την έκθεση Βάλιον θα δούμε άλλα δύο σημεία που έχουν να κάνουν με άλλες δύο εκθέσεις και θα έχουμε και την παρουσία των ε, των. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο σχετικά με την ημερήσια διάταξη, γι' αυτό ακριβώ περνάω στο σημείο 2. Παρακαλώ συνάδελφοι, έχετε μια κάποια αντίρρηση για τα πρακτικά της 20 Δεκεμβρίου 2011, 12 Ιανουαρίου 2012. 23 Ιανουαρίου 2012, καμία αντίρρηση, τότε εγκρίνονται τα πρακτικά των τριών αυτών συνεδριάσεων. Το σημείο 3 τώρα, ανακοινώσεις της Προέδρου. Αύριο το πρωί, στο τέλος της συνάντησης της Επιτροπής μας, Επισήμως θα δούμε μία αναφορά που προσυπέρεψαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες για τη Συμφωνία Άκτα και θα μας επιδοθεί αυτή η αναφορά εδώ μπροστά στην αίθουσα και θα γίνει παρουσία τύπου. Του τύπου λοιπόν ε, παρακαλώ όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να παραστούν αύριο μετά τις 12.30 να είναι εδώ. Τελευταία ανακοίνωση σας έχει δοθεί το παράρτημα στα φυλάδιο αυτό της Προεδρίας ε, και αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση τότε εγκρίνεται και αυτό το συνοδευτικό. Όχι, καμία αντίρρηση. αλλά λοιπόν, εγκρίνεται και το παράρτημα αυτό. Ξεκινάμε με το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, το θέμα για την γνωμοδότηση του κυρίου Σαλαβράκου για το 2013 που είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Σχετικά με την παρουσίαση των τροπολογιών προθεσμία μέχρι την 1η Μαρτίου του 2012, τρεχοντός έτος λοιπόν και η ψηφοφορία στην Επιτροπή στη συνάντηση της 20ης Μαρτίου. Ο κύριος Αλαβράκος έχει το λόγο για να μας κάνει την παρουσίαση λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, όπως σας είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το χαρακτηρισμό του έτους 2013 ως έτους των πολιτών. Το προτινόμενο ευρωπαϊκό έτος είναι χτισμένο από μια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 Τελικά μάλλον ήταν πρόβλημα μικροφώνου. Okay. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Σνάρφ. Ε, επαναλαμβάνω. Όπως είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το 2013 σαν Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Το προτινόμενο Ευρωπαϊκό Έτος είναι χτισμένο γύρω από μια ευρεία ενημερωτική εκστρατεία της Ένωσης. Ε, βεβαίως προσωπικά θα ήθελα να πω ότι κάθε χρόνο απομονώνουμε ορισμένες ωραίες ε, θεματικές πρωτοβουλίες τις χαρακτηρίζουμε σαν έτος των πολιτών και από εκεί και ύστερα μόλις περνάει το έτος έχει περάσει και η πρωτοβουλία και δεν έχουμε προχωρήσει σε ουσιαστικά ε, βήματα για να υλοποιήσουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν οι ωραίες πρωτοβουλίες τις οποίες κατά παίρνουμε. Και είναι γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών είναι όχι μόνο μία ε, πρωτοβουλία που θα μπορούσαμε να την πούμε συναισθηματική ή υψηλού επίπεδου από πλευράς αισθημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ουσιαστική διότι όπως καλά γνωρίζετε οι τελευταίες στατιστικές μας λένε ότι το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μια τεράστια μείωση του πληθυσμού, μια γύρανση του πληθυσμού και παράλληλα μια μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών οργών οι οποίοι θα κατοικήσουν τη χώρα πρέπει να ενσωματωθούν στις χώρες μέλη και εν γέννη στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους δούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τους εντάξουμε μέσα στις κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, προέρχομαι από μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία εκτός από τα οικονομικά της προβλήματα έχει μεγάλο πρόβλημα από λαθρομετανάστευση κυρίως όπως όλες οι άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, η Ιταλία, ε, η Γαλλία στην περιοχή της Μασαλίας της Μεσογειακής περιοχής η Ισπανία, η Πορτογαλία και θα πρέπει σαν μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας να δούμε το θέμα διότι χρησιμοποιούμε δυστυχώς την εργασία των ανθρώπων που προέρχονται από τις τρίτες χώρες και δεν, δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να τους ενσωματώσουμε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ε, Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε διάφορες απόψεις του θέματος. Ε, εγώ προέρχομαι από συντηρητικές απόψεις και από συντηρητική πολιτική ομάδα. Δεν πάω όμως να θεωρώ ότι τα προβλήματα και αν εναγκαλιστούμε τους μετανάστες τους οποίους ούτως ή άλλως θέλουμε δεν θέλουμε μας αρέσει ή δεν μας αρέσει θα τους έχουμε στις χώρες μας θα έχουμε κάνει μεγάλο λάθος. Ε, επομένως πρέπει όλους αυτούς στα πλαίσια της ενσωμάτωσης στην κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών να τους δώσουμε τη βελτίωση της επίγνωσης των δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη που θα τους επιτρέψει να παίρνουν συνειδητές αποφάσεις για το πώς θα ασκήσουν τα δικά τους δικαιώματα και πώς θα συμμετέχουν στην ελεύθερη κυκλοφορία τόσο των προσώπων όσο και των ιδεών και τον ισχυρότερο και τη δημιουργία ενός ισχυρότερου δεσμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της οι οποίοι 20 χρόνια μετά και θεωρώ ότι τα 20 χρόνια είναι πολιτικός χρόνος χθες είναι πολύ σύντομος πολιτικός χρόνος θα κληθούν να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνθρωποι μη προερχόμενοι από την Ευρώπη. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται σε ένα άλλο κράτο μέλος, κίνηση, το δικαίωμα αν κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος να ψηφίζουν και να είναι υποψήφοι στις τοπικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, δηλαδή στην Επιτροπή τη δική μας, το οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Αυτά είναι τα κύρια σημεία τα οποία προσπάθησα να καλύψω με την έκθεση και τις τροπολογίες μου. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ κάνοντας περαιτέρω ανάλυση ε, των τροπολογιών αφού μπορείτε να τις μελετήσετε θα ήθελα να σας παρακαλέσω οι όποιες τροπολογίες που κατερεθούν να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν στους στόχους της Επιτροπής της Επιτροπής Αναφορών και να μην ξεφύγουμε από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας αφού θα υπάρχουν και άλλες γνωμοδοτήσεις και άλλων επιτροπών ε, οι οποίες ε, θα καλύψουν το θέμα και ε, από μια γρήγορη ματιά που έριξα είδα ότι είναι αρκετά εμπεριστατωμένες και επαρκείς όπως και η έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Είμαι στην σα για οποιαδήποτε διευκρίνηση και θα δεχτώ με χαρά τι απόψει. Κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, εκείνο το οποίο θα ήθελα να σα πω, παρότι είμαστε λίγοι, είναι ότι τι τελευταίε εβδομάδε, λόγω και της οικονομική κρίση, παρουσιάζεται μια ρήξη των κοινωνιών των πολιτών στη βάση των λαών. Δηλαδή είχαμε το πρόβλημα οι Γερμανοί να υβρίζουν τους Έλληνες Γερμανοί πολίτες οι γερμανικές εφημερίδες να βρίζουν τους Έλληνες πολίτες, τους Ιταλούς πολίτες, οι Έλληνες με τη σειρά τους να βρίζουν τους Ιταλούς, να καίνουν γερμανικές σημαίες, να έχουν σβάστικα κτλ. κτλ. Αυτό με ενισχύει πάρα πολύ σαν πολιτικό, διότι θεωρώ ότι χωρίς να δημιουργείται καμία ουσιαστική επίλυση οποιοδήποτε θέματος που αναφύεται, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια στη βάση των λαών να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή συνείδηση πρέπει ε, η κρίση να περάσει πιστεύω ότι πολύ σύντομα ή αν δεν είναι σύντομα σε 4, 5, 10 χρόνια. Το θέμα είναι μετά να μην έχουμε διαρρήξει τις σχέσεις μας και να μπορούμε να κοιτάμε στοιχειοδός ο ένας τον άλλον και να μην έχουμε ανταλλάξει τέτοιες ύβρις σε επίπεδο λαών και σε επίπεδο προσώπων που θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα για τη μελλοντική επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα ο καθένας από εσά να προβληματιστεί πάνω στο θέμα και ίσως κυρία Πρόεδρε να δούμε σαν Επιτροπή Αναφορών διότι α, ε, ακριβώς η ρίζα η οποία δημιουργεί αυτά τα προβλήματα είναι η αγανάκτηση του μέσου πολίτη είτε του Έλληνα ο οποίος αισθάνεται να καταπιέζεται ή του, του Γερμανού που αισθάνεται ότι πληρώνει για τον Έλληνα ή τον Ιταλό ή οποιοδήποτε άλλο και να δείξουμε ότι πάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση και για μια Ευρωπαϊκή ιδέα συνενού των ανθρώπων όχι αναγκαστικά ανθρώπων οι οποίοι συμβιούν για ένα συμφέρον και μόνον διότι τα συμφέροντα όπως ξέρετε δεν είναι μενετά πολλές φορές αλλάζουν αυτό ήθελα να πω ευχαριστώ για τον χρόνο που μου αφιερώσατε και ε, ο προβληματισμός που σας έθεσα παρακαλώ να γίνει ουσιαστικότερος ευχαριστώ πολύ Κύριε Σαλαβράκο, σας ευχαριστούμε. Αυτά που μας είπατε, αυτά που μας είπατε σίγουρα θα αναλυθούν, θα εκτιμηθούν, θα γίνουν αντικείμενο σκέψεις για να δούμε ακριβώς εμείς τι κάνουμε για τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα και πολλές άλλες σκέψεις και συλλογισμοί υπάρχουν και θα πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε σας ευχαριστήσω ε, κύριε Σαλβαράκο για την παρουσίασή σας. Εξεπλάγιν λίγο, με την καλή έννοια. Γνωρίζω κάποιους από τους ε, συναδέρφους σας ε, στην πολιτική σας ομάδα. Δεν περίμενα μία θέση τόσο ανοιχτή όσο αυτή που παρουσιάσατε εδώ. Καταρχήν λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ για κάτι για το οποίο η Επιτροπή μας μπορεί να υπερηφανεύεται. Ε, εννοώ τη βάση για την έκθεσή σας. Δεύτερον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα των πολιτών να συμμετάσχουν. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ η διαφάνεια, η καλή διαχείριση, όλα τα πράγματα που χρειαζόμαστε στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι πολίτες μας να έχουν δυνατότητες, διότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα. Μερικές φορές όταν ακούω κάποια μέλη της Επιτροπής έχω την αίσθηση ότι πιστεύουν ότι στόχος είναι να προστατεύουμε την Κομισιόν από τους πολίτες και όχι να προστατεύουμε τους πολίτες όχι από την Επιτροπή, αλλά να προστατεύουμε τα δικαιώματα των πολιτών, να υπερασπιζόμαστε τη διαφάνεια. Θα κοιτάξουμε λοιπόν... Ε, θα θέλαμε να κοιτάξουμε και αυτό το σημείο, δηλαδή τη δυνατότητα συμμετοχής. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό και για την ένταξη των πολιτών, το να μπορούν να συμμετέχουν. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι νέο μέλος στην Επιτροπή από την αρχή του, αυτού του χρόνου. Θα ήθελα να πω δύο λόγια. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια. Πρόεδρε, συγχωρέστε με αν είμαι ακριβώς μέσα στο θέμα ή στο πνεύμα των συζητήσεων. Ελπίζω να είμαι. Αν η συνάδελφος εξεπλάγει μια φορά από τη γνωμάτευση του κυρίου Σαλαβράκου, εγώ ως Έλληνας και ανήκοντας σε διαφορετικό διαμετρικά πολιτικό χώρο είμαι εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ εξεπλάγει δυο φορές θετικά ο κύριος Σαλαβράκος με τις βασικές παρατηρήσεις και τις τροπολογίες ε, είμαι σύμφωνος υπερεύει σε βασικά σημεία τις συντηρητικές παραδόσεις όπως μας είπε ο ίδιος του χώρου του. Επιτρέψτε μου να πω ότι πρόκειται περί μιας αξιόλογης προσπάθειας του κυρίου συναδέλφου αλλά πρόκειται περί ενός προβληματισμού που ανέπτυξε και στο οποίο αναφέρεται η σχετική ε, γνωμοδότηση η οποία μας αφορά όλους που σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε ορισμένες προδιαγραφές πώς βλέπουμε τα δικαιώματα των πολιτών στην Ευρώπη. Πρώτον, είναι υποκριτικό να ανακηρύσσονται έτοιμοι κατά τη φτώχειας και η φτώχεια να μεγαλώνει κατά της ανεργίας και η ανεργία να μεγαλώνει και φέτος να πούμε έτος των πολιτών και τα δικαιώματα των πολιτών να περιορίζονται. Αυτό δεν είναι λογοτεχνικό σχήμα. Πιστεύω ότι η κρίση οικονομική που μαστίζει την Ευρώπη και την Ελλάδα δεν είναι μόνο κρίση οικονομική. Είναι κρίση δημοκρατίας, άρα κρίση των δικαιωμάτων των πολιτών. Και προβλέπω κυρία Πρόεδρο και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, ότι θα έχουμε στο έτος κατά τα άλλα των δικαιωμάτων των πολιτών πάρα πολλές αναφορές από πολίτες όλης της Ευρώπης ενδεχομένως τα στατιστικά να πούν από πολίτες των χωρών της Νότιας Ευρώπης που θα απευθύνονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα απευθύνονται σε μας με βασικό αντικείμενο Το μικρόφωνο σας, το μικρόφωνο σας. Το μικρόφωνο σας η γνωμάτευση του κυρίου Σαλαβράκου είναι μια καλή υποδοχή το τι μας περιμένει τον επόμενο χρόνο. Με αυτή την έννοια αυτά ήθελα να πω, συμφωνώ με τις βασικές παρατηρήσεις και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια σωστή γνωμοδότηση και να βοηθήσουμε όσα είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι και όσα και εγώ ως νέο μέλος προσπαθήσω να κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τζανόκα. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σε χαρώ τον κύριο Σαλαβράκο ε, για τις ε, απόψεις, και τις ε, απόψεις του και τις ιδέες του. Ορισμένες από αυτές φαντάζομαι δεν ε, βρίσκουν σύμφωνους ε, ορισμένου συναδέλφου από αυτήν τη συγκεκριμένη πολιτική ομάδα. Πολύ πρόσφατα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ψηφίστηκε η, γνωμοδο... η έκθεσή μου η γνωμοδότησή μου για την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την την για το 2010 και οι συνάδελφοι από τη στηρητική ομάδα και το ΕΛΚ ήταν αντίθετοι με ορισμένε από τι θέσει που αναφέρατε και εσεί στη δική σα ε, γνωμοδότηση, ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των ε, πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνάδελφοι ήταν ε, αντίθετοι με την θέση μου, ακόμα και σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων των ε, κατοίκων και των πολιτών, δηλαδή των ατόμων που διαμένουν απλώ και των πολιτών. Εσεί αναφερθήκατε στο δικαίωμα της ελεύθερη ε, κυκλοφορία. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί αυτή τη στιγμή μόνο στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στον κανονισμό θεωρήσεων και δεν συμπεριλαμβάνεται η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ξέρετε. Επομένω, εκεί δεν μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Βεβαίω, εμεί θα θέλαμε και στηρίζουμε απολύτω το ενδεχόμενο να είναι δυνατή άσκηση του δικαιώματο ε, στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Συμφωνούμε απολύτω λοιπόν. Πρέπει όμως να εργαστούμε από αυτών των ζητημάτων. Και στο πλαίσιο όλων αυτών των συζητήσεων για την ε, κοινωνική ενσωμάτωση έχουμε θίξει και αυτό το ζήτημα. Ακόμα και όσοι έχουν ε, άδεια παραμονής, ή και οι απάτριδες ε, πολλές φορές αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Ακόμα δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερη κυκλοφορία ε, στην Ιρλανδία και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Συζητήσαμε την έκθεση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εγώ είμαι μέλο αυτή τη Επιτροπή. Ε, συμφωνούμε, στηρίζουμε την ε, πρόταση αλλαγή του τίτλου της έκθεσης. Να μην αποκαλείται έκθεση για τους πολίτες, citizens, αλλά citizenship. Για την ηθαγένεια. Γιατί δίνεται η εντύπωση ότι υπογραμμίζουμε τη σημασία της ηθαγένειας ως θέματος που χορηγεί δικαιώματα ε, στους ε, πολίτες που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την ιδέα ή όχι, αλλά στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ο εισηγητής και η πλειονότητα των ε, συναδέλφων ε, υποστήριξε αυτή την ιδέα αλλαγής ε, του τίτλου για να τονίσουμε ότι μιλάμε εδώ για την ηθαγένεια που είναι ένα από τα χαρακτηριστικό των δικαιώματων των οποίων χαίρουν όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι πολίτες το κατά πόσο δηλαδή τους ε, εγχωρούμε ορισμένα δικαιώματα. Ίσα δικαιώματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παναλαμβάνω λοιπόν ότι η ομάδα μας ε, νομίζω θα στηρίξει ε, τις προτάσεις σας και ενδεχομένως να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Γενικώ πώς όμως συμφωνούμε με την έκθεσή σας. Έχω, μπερδευτεί λίγο. Έχουμε ε, προχωρήσει στη συζήτηση ή ακούμε τους σκιώδες συζητητές. Σε ποια φάση βρισκόμαστε. Είναι ανοιχτή η συζήτηση. Διότι σε άλλες ε, ομάδες πρώτα ακούμε ε, την παρουσίαση της έκθεσης και μετά τους, ε, ακούμε τους κύριους συζητητές. Ε, εντάξει, εγώ θα πω τη γνώμη μου λοιπόν ε, ως ε, σκιώδης εάν μου επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ, λέει η πρόεδρος. Η ακούμε τη συζήτηση μεταξύ των ε, Ελλήνων συναδέρφων και ήταν πολύ ενδιαφέρον που ε, τέθηκε σε πιο ευρία βάση το θέμα. Δεν μιλάμε μόνο για το ίδιο το έγγραφο, μιλάμε και για ε, τις επιδράσεις και τις διαδικασίες που υπάρχουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε λοιπόν για το θέμα των πολιτών, το έχουμε συζητήσει και στα πλαίσια της ΑΚΤΑ. Χθες ε, λοιπόν υπήρχε σαφές ε, πνεύμα πολιτών ε, από πλευράς των πολιτών μας. Ποτέ δεν έλαβα τόσα email, τόσα ηλεκτρονικά μηνύματα που να ξεκινούν εγώ ως Ευρωπαίος πολίτης. όλα αυτά στα πλαίσια της συζήτησης για, για την νομοθεσία ΑΚΤΑ. Η συζήτησή μας θα πρέπει στόχο να έχει να ενισχύσει το πνεύμα των ε, πολιτών. Ε, και μάλιστα ως θετική ιδιότητα, όχι μόνο ε, όταν κινητοποιούνται οι πολίτες ενάντια σε κάτι, όπως στην περίπτωση της νομοθεσίας Άκτα. Η έκθεση αυτή, η γνωμοδότηση αυτή μιλά για την ελευθερία κίνησης και θα ήθελα για την ελεύθερη κινητικότητα και ένα ζωτικό θέμα που θα ήθελα να προσθέσω στις τροπολογίες μου είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών ε, πριν τις ευρωεκλογές, διότι δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στην ελεύθερη κινητικότητα. Θα πρέπει επίσης, όπως είπα, να δημιουργήσουμε ένα θετικό πνεύμα ε, μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. κατά τις εκλογές, ε, τις τοπικές, ε, τις εθνικές και τις ε, ευρωεκλογές. Θα πρέπει λοιπόν να προσθέσουμε κάποιες τροπολογίες και που αφορούν τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και στα εκτιμώντας και στο διατακτικό του κειμένου. Οι, ευρωπαϊκοί, οι ευρωπαίοι πολίτες θα, πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να προστατεύονται από τις ε, διπλωματικέ αποστολές τη Ευρωπαϊκής Ένωση σε τρίτες χώρες. Και αυτό είναι δικαίωμα των πολιτών μας. Όπου και να πάνε λοιπόν, όταν μιλάμε για ελεύθερη κινητικότητα, συνήθως μιλάμε για ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όμως και οι πολίτες μας να προστατεύονται από τις πρεσβείες και τις αποστολές μας εκτός της Ευρώπης. Επίσης, πιστεύω ότι Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε και να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τον ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή καθώς και της ε, Επιτροπής μας, της Επιτροπής των Αναφορών. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να γνωρίζουν το γεγονός ότι παίζουμε σημαντικό ρόλο ε, απαντώντας ε, στις ε, ανάγκες, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις ελπίδες των πολιτών μας. Ελπίζω λοιπόν στο άρθρο 4 να ρυθμίσουμε το θέμα του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 4 λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά ε, τα μέτρα που υπάρχουν στο παράρτημα. Ε, θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ κάποια πράγματα. Αυτά θα είναι τα βασικά στοιχεία που πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε στις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Έλμερ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σκεφτόμουν ότι η Ευρωπαίοι πολίτες και Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα ήθελαν να γνωρίζουν ότι εδώ στις Βρυξέλλες έχουμε μάτι υψηλά αμοιβόμενους ανθρώπους που φαίνεται να συζητούν αν θα πρέπει να έχουμε Ευρωπαϊκό έτος πολιτών ή Ευρωπαϊκό έτος ε, Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Ε, Νομίζω ότι πολλοί πολίτες ε, θα θεωρούσαν ότι είναι καλά τα τα χρήματα αυτά, αναρωτιέμαι. Βρίσκομαι Είμαι μέλος και της Επιτροπής ε, Απασχόλησης και έχουμε συζητήσει εδώ πολλά, προβλη... πολλά προγράμματα όπως είναι το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων ή το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρανσης. Ε, αυτά, ενεργού γύρανσης. Αυτά ε, μας απασχολούν εδώ ως βουλευτές, ε, τα συζητάμε επί μακρόν και ε, τολμώ να πω ότι κανένας από τους πολίτες στα κράτη-μέλη μας ούτε έχουν ακούσει αυτές τις πρωτοβουλίες, ούτε έχουν επαφεληθεί από αυτές, ούτε και τους νοιάζει πολύ. Και υποψιάζομαι ότι σε μεγάλο βαθμό το ίδιο θα ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, σήμερα, μέχρι σήμερα δεν είχα ακούσει τίποτα για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών και τολμώ να στοιχηματίσω ότι όταν περάσει αυτή η χρονιά και ε, όταν θα την κοιτάμε αναδρομικά, σχεδόν κανένας πολίτης δεν θα έχει ακούσει από το έτος αυτό, ε, ούτε θα έχει αποφεληθεί από αυτό. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί το κάνουμε. Κάποιες από τους παραλύσαντες πολύ σωστά ε, επέστησε την προσοχή μας σε μια κρίση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν σκεφτούμε ποια είναι τα δικαιώματα του πολίτη, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μεταξύ άλλων το δικαίωμα του εκλέγην και τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή έχουν αρχηγούς κυβερνήσεων που τους έχουν επιβληθεί από τις Βρυξέλλες, τους οποίους δεν ψήφισαν. Στην περίπτωση της Ελλάδας ε, όλες οι δημοσκοπήσεις ε, φαίνεται να δείχνουν ότι θα ψηφίσουν κάποιο τελείως διαφορετικό. Μπορεί να, λοιπόν, να λέμε ότι θέλουμε για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν επιτρέπουμε στον κόσμο να εκλέγει τους πολιτικούς ηγέτες τους. Και ε, υποψιάζομαι ότι αν κάποιοι από τους εργάτες ή μη εργαζομένους από τους δρόμους των Αθηνών εδώ μπορεί να μιλούσαν για το δικαίωμα στην απασχόληση και το δικαίωμα αξιοπρεπούς πληρωμής, τέτοια πράγματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πολύ περίεργη θέση. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολύ σημαντική κρίση. Κάποια κράτη-μέλη βρίσκονται σε πολύ δύσκολες ε, περιστάσεις και αυτή τη στιγμή μιλάμε για ε, το ε, για, για, για, τα δικαιώματα του πολίτη που μάλλον δεν ενδιαφέρουν και πολλοί αυτούς που καίνε ευρωπαϊκές και γερμανικές ε, σημαίες στην, ε, στους δρόμους των Αθηνών. Και τι ακριβώς είναι το πνεύμα του πολίτη. Εγώ εκπροσωπώ 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και αν τους ρωτήσω ε, είσαστε πολίτες τίνος, μερικοί θα λέγανε της Αγγλίας, μερικοί θα λέγανε του Ηνωμένου Βασιλείου, μερικοί θα λέγανε της Μεγάλης Βρετανίας. Νομίζω ότι ούτε 1% δεν θα έλεγε ότι είμαι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάποια έννοια με νόημα. Μπορεί λοιπόν να λέμε εδώ πέρα ότι θέλουμε, μπορούμε να δημιουργούμε προγράμματα, μπορούμε να ε, περνάμε το χρόνο μας ε, δημιουργικά και να είμαστε περήφανοι για τόσα όσα έχουμε κάνει, αλλά η δική μου ανησυχία είναι ότι αυτό δεν θα κάνει καμία διαφορά για τους ανθρώπους ε, των οποίων τη ζωή θέλουμε να επηρεάσουμε. Και εκείνοι μάλλον θα πιστεύουν ότι μπορούμε να περάσουμε το χρόνο μας πολύ πιο επικοδομητικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Χέφνερ τώρα. Χέφνερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να οριστεί αυτό το έτος ως έτος Ευρωπαίων Πολιτών και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την πρόταση της Επιτροπής. Αλλά πρέπει να δούμε να καταλάβουμε ότι αν δεν έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που προτείνονται στην ε, γνωμοδότηση, προφανώς δεν έχουμε αξιοποιήσει στο έπακρον. Επιτρέψτε να μιλήσω στα γερμανικά. Αν πραγματικά θέλουμε ένα έτος των πολιτών, και αν δεν θέλουμε να συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα, business as usual, τότε η χρονιά αυτή θα είναι κάτι παραπάνω από μια ευκαιρία να πούμε στους πολίτες πόσο καλή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πόσο καλά λειτουργεί και τι δικαιώματα έχουν. Όλα αυτά είναι σημαντικά ε, και αναφέρονται στην πρόταση. Εγώ θα ήθελα να προτείνω ακριβώ εδώ στην Επιτροπή Αναφορών το θέμα μήπως το έτος πολιτών θα πρέπει να είναι έτος κατά το οποίο οι πολίτες ε, της Ευρώπης να νιώσουν ότι τους παίρνουμε στα σοβαρά και ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινή Ευρώπης. Το θέμα δηλαδή δεν είναι μονομερός να επικοινωνούμε από την πλευρά των θεσμικών οργάνων προς τους πολίτες, αλλά ε, αντίστροφα θα μπορούσαμε να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες των πολιτών από την Ένωση, ποιες είναι οι προτάσεις τους. Δηλαδή, ε, αυτή τη χρονιά να πάρουμε πιο σοβαρά τι δυνατότητε συμμετοχή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι κάνουμε συνήθω και να υποβάλουμε σχετικέ προτάσει. Ένα στοιχείο είναι το 2013. θα εφαρμοστεί πρώτη φορά πραγματικά η ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ε, τον Απρίλιο ξεκινάει, αλλά μέχρι η Πρωτοβουλία των Πολιτών ε, μέχρι πρωτοβουλίες των πολιτών ε, να ε, ολοκληρωθούν, να συγκεντρωθούν οι υπογραφές, ε, να γίνουν οι διαβουλεύσεις. Θα έχουμε φτάσει στα τέλη του 2012, αρχές του 2013. Και πιστεύω ότι καλό θα είναι σε, κατά διάρκεια αυτού του έτους των πολιτών να έχουμε κατά νου να ενισχύσουμε το στοιχείο αυτό, να καλέσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από το δικαίωμα αυτό, από τους οποίους πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεύτερον, θα ήθελα τη χρονιά αυτή να την ε, εκμεταλλευτούμε ώστε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με τους πολίτες, να ακούσουμε ποιες είναι οι προσδοκίες τους ε, και να έχουμε έναν μόνιμο διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό ήθελα να προτείνω και βλέπω την Επιτροπή μας ως την Επιτροπή που ε, ακριβώς ασκεί αυτό το καθήκον ε, ε, στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να περιλάβουμε το στοιχείο αυτό στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Προσθέτοντας ή απαντώντα στον συνάδελφο Χέφνερ, θα ήθελα ε, να πω και εγώ κάτι. Εγώ είμαι υπέρ ε, του προγράμματος αυτού. Ε, θα μπορούσε να το διατυπώσει κανείς διαφορετικά. Φυσικά υπάρχουν ελλείμματα και στην πολιτική θα πρέπει να αναλαμβάνει κανείς ε, ηγετική θέση. Ε, είδαμε ότι μετά τους ε, παγκοσμίους πολέμους είδαμε ειρηνικές εποχές στην Ευρώπη, είδαμε ότι το σιδηρούν παραπέτασμα έπεσε, είδαμε και την επανένωση της Γερμανίας. Το έλλειμμα έγκυται στο ότι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις τις οποίες πολύ σωστά έχει λάβει η ελίτ, θα πρέπει ε, να μεταφερθούν στους πολίτες και οι πολίτες να συμμετάσχουν ε, στην Ευρώπη και να ενταχθούν ε, στην Ευρώπη. Ο ίδιος πολίτης, και υπάρχει εδώ μια αντίφαση, ο πολίτης που επικρίνει έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτόν τον πολίτη θα μπορούσαμε να του πούμε φαντάσου ότι δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, από εκεί που μένω εγώ, ε, σε μισή ώρα ε, φτάνει κανείς στα σύνορα. Θα έπρεπε λοιπόν κανείς να περιμένει στα σύνορα, να φοβάται με τα σύνορα αυτά έχανε κανείς τα δικαιώματά του, εξαρτιόταν κανείς από τα καπρίτσια ενός τελωνιακού. εγώ λοιπόν Σας καλώ το έτος των πολιτών ε, να το ε, κάνουμε κατανοητό για τους πολίτες, γιατί είναι κάτι που χρειάζονται. Να το πω διαφορετικά. Εάν δεν πετύχει τώρα αυτό, το πρώτο βήμα ήταν καλό, ήταν σωστό. Ε, ε, μετά, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η πολιτική ελίτ ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όμως ε, θα πρέπει αυτό το εγχείρημα να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε στο κάθε άτομο. Εάν αυτό αποτύχει τότε θα αποτύχει όλο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των πολιτών. Αυτά εισαγωγικά διότι βρίσκω πολύ χρήσιμη και ε, ε, και, και λογική μια τέτοια πρωτοβουλία. Ε, οι πολίτες είναι οι πολίτες ε, είναι το περιβάλλον από το οποίο θα βγουν όλα αυτά και ε, η, Ευρωπαϊκή, η Ελλάδα διαμαρτύρεται επειδή ε, νιώθει ότι δεν την καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να λάβουν βοήθεια όχι ως ελεημοσύνη αλλά βοήθεια για να τα καταφέρουν μόνοι τους. Αυτό ήθελα να πω. Όσον αφορά την ίδια την έκθεση, θα πρέπει να την διαβάσουμε αναλυτικά. Ε, εμένα ε, με απασχολεί το εξής. Ε, υπάρχουν κάποια δικαιώματα, αλλά δεν θα πρέπει να εξετάσουμε και τις, τις υποχρεώσεις, διότι εγώ ως πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης έχω όχι μόνο δικαιώματα, έχω και υποχρεώσεις. Ε, αναφέρατε και την ένταξη των μεταναστών. Ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα. Ε, πολύ σωστά το ανέφερε αυτό ο συνάδελφος Σαλαβράκος. Ε, χρειαζόμαστε ε, την ε, μετανάστευση στην Ευρώπη διότι λόγω των δημογραφικών εξελίξεων θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε προσπάθειες για την ένταξη των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστώ. Τώρα αν δεν έχουμε κάποια άλλη παρέμβαση, νομίζω ότι και αυτό συμβαίνει. Ο κύριος Σαλαβράκος και πάλι έχει το λόγο, μήπως θα ήθελε να μας πει κάτι καταληκτικά. Ε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την τοποθέτηση, ε, θετική τοποθέτηση πάνω στην έκθεση και ήθελα να μοιραστώ τον εξή προβληματισμό. Όταν μιλάμε για οικονομία, όταν ε, σπούδαζα οικονομικά, ε, τι είναι οικονομία έλεγε ο καθηγητής μου, expectation τι είναι πολιτική expectation, τι είναι ζωή expectation. Δεν είναι desire. Ε, αν φιλολογικά έχει διαβάσει κανείς τόσα παίρνει ο άνεμος, κλείνει με το αύριο θα είναι μια άλλη μέρα. Αυτό τι δείχνει. Expectation. Το θέμα είναι αυτή την expectation, αυτή την προσδοκία, να μην την κόψουμε από τους πολίτες. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των πολιτών. Απόλυτα. Αλλά θα προσπαθήσουμε και τουλάχιστον να τους το υποδείξουμε. Δηλαδή συμμερίζομαι του κυρίου Έλμερ τις ανησυχίες ε, για τη ρεαλιστικότητα αλλά δεν μπορούμε να κόψουμε και τη φαντασία του ανθρώπου. Πρέπει να ζούμε ε, σε μία ε, ρεαλιστική, ό, ό, όχι ένα virtual reality, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια ρεαλιστικη οχι ενα virtual reality αλλα εν παση περιπτωσει σε μια προσδοκια σε expectation. Αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω και όσον αφορά το θέμα ηθαγένεια έχουμε προβλήματα όπως ξέρετε με το Δουβλίνο, Δουβλίνο 2. Πρέπει να το δούμε. Εδώ πρέπει να δώσουμε τη γραμμή ακριβώς της ευχής να γίνουν ορισμένες μεταβολές σε θέμα με το distribution των μεταναστών, διότι έχουμε το distribution των μεταναστών από το 2, που δεν είναι αντικείμενο της παρούσης εκθέσεως. Ο προβληματισμός τίθεται όμως στην έκθεση αυτή, γιατί διότι θα αναγκαστούμε σε 10-20 χρόνια να προσαρμοστούμε σε μια νέα κατάσταση. Και όπως λένε οι φίλοι μας οι Βλέζοι, δεν θέλω να ε, έχουμε την παροιμία ε, όταν έχεις έναν βιασμό και δεν μπορείς να τον αποφύγεις απόλαυσέ τον. Θέλω να αποφύγω το βιασμό. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και αυτό προσπαθώ με την έκθεση να δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Σαλαβράκο, όπως επίσης και τους κοιόδες εισηγητές. Κλείνουμε το σημείο αυτό. Προθεσμία και τις τροπολογίες 1η Μαρτίου. Το επόμενο σημείο τώρα της ημερήσιας διάταξης έχει να κάνει με περίπου 26 αναφορές που υπέβαλαν πολίτες της περιοχής της Καμπανία στην Ιταλία για τη δυσκολία για τα απόβλητα στην Καμπανία και την κατάσταση αυτή την παρακολουθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα η Επιτροπή μας ε, από το Δεκέμβριο του 2009 και τότε ακριβώς ε, είχαμε αρκετούς πολίτες από την Καμπανία που είχαν προσυπογράψει διάφορες τροπολογίες, ε, συγγνώμη, αναφορές και παρακολουθήσαμε έτσι την όλη πορεία που οδήγησε την ε, περιφέρεια της Καμπανίας επιτέλους να υιοθετήσει συγκεκριμένο σχέδιο και πρόγραμμα για τα απόβλητα και να το υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή του σχεδίου αυτού. Ακούμε όμως και άλλες παρατηρήσεις από πλευράς πολιτών για την νομιμότητα του προγράμματος του σχεδίου αυτού αν ε, είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αν θα πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό όπως έχει προταθεί και αν συμφωνεί με όλα αυτά που ισχύουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι ότι μείωσε την προστασία η Επιτροπή πριν από δέκα περίπου μέρες να σας πούμε ότι είχε στείλει αντιπροσώπους της ε, στην Καμπανία, στην Ιταλία για να δει πως έχει κατάσταση. Άρα λοιπόν ε, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και πάλι οπωσδήποτε να καλέσουμε αυτές τις αρχές για να μας δώσουν τη δυνατότητα να ακούσουμε όπως επίσης και στους πολίτες του Ιταλούς της Καμπανίας για όλα αυτά που συμβαίνουν και να τους ε, ε, καθησυχάσουν ε, ότι το σχέδιο αυτό αποτελεί πραγματικά μία λύση. Ανέφερα διάφορα ονόματα, θα λάβουν όλοι το λόγο με παρεμβάσεις, αλλά σας παρακαλώ να σεβαστείτε τα όσα σας έχουμε διανύμει και ακριβώς από τον Περιφερικό συντονισμό για τα απόβλητα της ε, καμπανίας Ζαμπιέρο Άντζελη, εκπρόσωπο Επιτροπής Επιτροπών, το Μάζο Εσπόζητο επίσης που εκπροσωπεί στην Ατσέρα τους πολίτες, όπως επίσης επειδή και διάφορες απουσίες, τις παρατηρήσεις του Τομάδο Σοντάνο από την Άπολη που είναι και γερουσιαστής και μας έστειλε γραπτά τις παρατηρήσεις του επειδή αδυνατή να παραστεί. Ο Δ. Ραϊμόντο Σαντακρότσε, συντονιστή όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή τη Καμπανία, για να μα κάνει την εισήγησή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν σας κρύβω τη συγκίνησή μου που μετά από δύο χρόνια επιστρέφω στην αίθουσα αυτή για να σας εξιστορήσω τα όσα κάναμε αυτά τα δύο χρόνια ακριβώς. Το σημαντικότερο, η σημαντικότερη μας ενέργεια ήταν να εγκρίνουμε το περιφερειακό πρόγραμμα αστικών αποβλήτων αυτό εξετάστηκε και κρίθηκε θετικά και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, εκτός από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και η Περιφέρεια από όταν ε, έπαυσε η διαχείριση περιφερειακή, τότε όταν είχαμε έρθει εμείς εδώ, ολοκληρωνόταν αυτή η φάση, και εγκρίθηκε επίσης το ειδικό πρόγραμμα αποβλήτων που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εγκριθεί και από το Συμβούλιο της Περιφέρειας της Καμπανίας. Και όπως ανακοινώσατε, έχει ενημερωθεί η Επιτροπή και χρειάζεται οπωσδήποτε να τονίσουμε το ότι οι διάφορες διαδικασίες μετά από τα σχέδια αυτά νομίζουμε ότι συμβαδίζουν με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Να ανοίξω μια σύντομη παρένθεση εγκρίναμε και το πρόγραμμα εξυγίανσης που λόγω του περιοχικού προγράμματος ακριβώς είναι από τα μέρη τα ουσιαστικά τα κύρια του συνολικού προγράμματος διαχείρισης των αποβλήτων. Το... Η πτυχή εξυγίανση λοιπόν. Άρα λοιπόν από διαδικαστικής πλευράς ακολουθήσαμε το σωστό δρόμο και ιδιαίτερα προσέξαμε την φάση την ε, δημόσια και όπως προβλέπει και η οδηγία για την εκτίμηση του πώς επί αποστατικής πλευράς επίσης ε, και ακολουθήσαμε τις τακτικές διαδικασίες ε, δημοσίου του scoping πριν από τη σύνταξη του σχεδίου ακριβώς για να έχουμε όλα τα στοιχεία από τους κοινωνικούς εταίρους όπως επίσης και τους φορείς που έχουν αρμοδιότητες για το περιβάλλον και το πώς συνδυάζονται τώρα αυτές οι ρυθμίσεις και πώς υπάρχουν παρεμβάσεις και συνδυασμοί με άλλα σχέδια και προγράμματα της περιοχής. Και μετά από τη σύνταξη του σχεδίου το υποβάλαμε προς εξέταση, το δημοσιεύσαμε και είχαμε και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να γίνουν παρατηρήσεις. Εξετάσαμε, προσφέραμε απαντήσεις στην έκθεση περί περιβάλλοντος και απαντήσαμε σε όλες τις παρατηρήσεις που μας έγιναν και μετά βάση του συνόλου της εργασίας μας ε, ακούσαμε και την γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα για αυτή την στρατηγική εκτίμηση και μόνο μετά από όλα αυτά πήγε αυτό στο Συμβούλιο το αρμόδιο και εγκρίθηκε. Και μετά από όλα αυτά να σας θυμίσω ότι στην περιφέρεια η περιφέρεια θα πρέπει να σεβαστεί τον προγραμματισμό. Άρα λοιπόν κατευθυντής γραμμές στις ε, τοπικές αρχές και ακριβώς ε, μετά από την έγκριση αυτή ξεκινήσαμε, μάλλον πριν από την έγκριση αυτή, ξεκινήσαμε διαβουλεύσεις και επίσημες διαβουλεύσεις με τις ε, επαρχιακές διοικήσεις ώστε να προσδιορίσουμε λεπτομεριακά μάλιστα ποια χρονική στιγμή αυτά θα πρέπει να γίνουν, όπως επίσης και τι επιλογές πρέπει να γίνουν σχετικά με το πού αυτά θα εγκατασταθούν. Και επίσης, συμπληρώντας όλα αυτά, οι χρηματοδοτήσεις. Γιατί η Ιταλική κυβέρνηση από τη στιγμή που δεν υπάρχουν περιφερειακές χρηματοδοτήσεις, ε, θα το γνωρίζετε ότι ε, δεν μπορούν ε, να χορηγηθούν μετά από απόφαση περιφερειακή. Τελικά δόθηκαν 150 εκατομμύρια ευρώ για να ενδυναμωθεί οι ενέργειες αυτές και να μπορέσουν να εγκατασταθούν νέοι μηχανισμοί και αυτό το σχέδιο για τα αστικά κυρίως απόβλητα, αυτό μας απασχολεί, αυτό μας αφορά, αυτό που επηρεάζει περισσότερο την περιοχή αυτή, επειδή δεν υπάρχει μια οριζόντια στρατηγική και προβλέπονται εδώ εγκαταστάσεις αποτέφρωσης και μάλιστα έχουμε και ενέργεια που κερδίζουμε και επίσης προβλέπονται σε ορισμένες περιπτώσεις και μάλιστα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή εγκαταστάσεις που ε, ε, συμπίκνωσης ε, με μια κατάλληλη συλλογή. Και επίσης χάρη στα χρήματα αυτά από πλευράς κυβέρνησης βέβαια θα δούμε και το τι λεφτά οφείλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινήσαμε και σχεδόν ολοκληρώσαμε α, τρεις εγκαταστάσεις, δύο στο Σαλέρνο και μία στην Καζέρτα για την κομποστοποίηση αυτών των προϊόντων. Και αυτό το τελευταίο θα ανοίξει, α, μάλλον ένα τέταρτο θα ανοίξει σε λίγους μήνες. Έχουν προωθηθεί εργασίες και όπως και η οι εκπρόσωποι από την επαρχία του Σαλέρνο θα μπορούσαν να, να μας αναλύσουν στη συνέχεια. Στην Καμπανία έχουμε ένα αποτεφρωτή στην Ατσέρα στη... και είχαμε την επίσκεψη της Επιτροπής στην Ατσέρα, στις εγκαταστάσεις εκεί, όπως επίσης ε, και στο θάλαμο που γίνεται ο σχετικός έλεγχος, η καθοδήγηση και δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω έχουμε μόνο στα Ιταλικά και μπορούμε να πάτε στο παρατηρητήριο περιβάλλοντος ε, της Ατσέρα και εκεί βλέπετε τις μετρήσεις της εκπομπές στην ε, ατμόσφαιρα μόλις την προηγούμενη μέρα. Και αν θέλετε έχω και ένα αντίγραφο εδώ που έχω τυπώσει σχετικά με το πώς κερδίζουμε, παίρνουμε ενέργεια η επαρχία του Σαλέρνο προκήρυξε το διαγωνισμό για ένα δικό τους αποτεφρωτή και υποκειμενικά και από το πως έχει ροή των πραγμάτων και σαν επίτροπο σχετικής επιτροπής ανάθεσης να σας πω ότι αυτό το σχέδιο όπως προκηρύχθηκε από το Σαλέρνο ε, ζητάει την καλύτερη τεχνολογία για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και τον πώς θα μπορούν έτσι να ελεγχθούν οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα οι καλύτερες δυνατές μέθοδοι και επίσης προβλέπονται πάντα στην επαρχία του Σαλέρνο κάτι που χρειάζεται να υπενθυμίσω είναι ότι ήδη λειτουργεί εκτός από τις τρεις αυτές εγκαταστάσεις μία στην Καζέρτα, δύο στο Σαλέρνο έχουμε και ε, με βιοαν διαδικασία με, σε, με αναεροβική μέθοδο. Έχουμε μια σχετική εγκατάσταση που ολοκληρώνεται τώρα. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία που χρησιμοποιεί μέθοδο αναεροβική έχουμε εγκαταστάσεις που διαχωρίζουν ε, τα απόβλητα με ένα ειδικό όνομα. Δεν ξέρω αν τα επισκεφθήκατε όταν πήγατε εκεί. Αλλά στις εγκαταστάσεις αυτές θα έχουμε ακριβώς ε, ζωντανούς οργανισμούς που θα αφομοιώνουν βιολογικά αυτά τα απόβλητα ε, και έτσι με οργανικό τρόπο θα παράγουν ενέργεια και αυτό όσον αφορά την επεξεργασία των αποβλήτων. Να σας πω ότι με τις χρηματοδοτήσεις που σας λέγαμε ασχοληθήκαμε και πάλι με το πώς θα έχουμε μια διαφοροποιημένη συλλογή σε συνεργασία με τους Δήμους και μέσω των επαρχιών που με το Υπουργείο Περιβάλλοντος έκλεισαν μια συμφωνία περιφέρεια της ε, Καμπανίας και ε, με μαζί με όσους έχουν ε, το αμπαλάζ, το περιτύλιγμα, το περίβλημα, μια συμφωνία βάση ενός προγράμματος με το, με το σχετικό φορέα για το περίβλημα. Στην καμπανία έχουμε ακριβώς ε, την επιτυχία αυτού του προγράμματος για μια διαφοροποιημένη συλλογή και ο έλεγχος είναι συγκεκριμένος ε, για τη συλλογή σε όλους τους δήμους αποβλήτων γιατί έχουμε με, με περιφερειακό νόμο ε, τα έχουμε προσδιορίσει αυτά βλέπουμε τι γίνεται με τον κάθε Δήμο και με την τοπική διοίκηση που συναντιούνται. Αναπτύξαμε προγράμματα για να βοηθήσουμε τους Δήμους εκεί που ισχύει αυτή η διαφοροποιημένη συλλογή ε, αλλά χωρίς καλό θετικό αποτέλεσμα. Και κάτι το τελευταίο, α, μισό λεπτό, εκπρόσωποι της περιφέρειας θα μπορούσαν να λάβουν το λόγο, αλλά το σημαντικό είναι να σας πω ότι ξεκινήσαμε και τη σύνταξη ενός ε, προγράμματος ελαχιστοποίησης των αποβλήτων και εγώ ίδιος με πόρους της περιφερειακής διοίκησης εδώ έχω προβλέψει την χρηματοδότηση με 6 εκατομμύρια ευρώ υπέρ των επαρχιών της Καμπανίας οι αδράσεις ελαχιστοποίησης αποβλήτων. Τι σημαίνει αυτό. Εδώ λοιπόν να δούμε πώς θα συμπυκνωθούν και αποχρωτικές περιοχές, πώς ε, Ε, με τα απορριπαντικά, τη χρήση τους σε συλλογική χρήση όπως σε σχολεία εδώ εκεί και πώς θα δώσουμε κίνητρα μέσω κατάλληλου ύδατος ε, φιλτραρισμένου εκεί που θέλουν ένα απόλυτα σίγουροι οι πολίτες ότι το νερό που πίνουν δεν είναι μολυσμένο αλλά εντάξει, να μην είναι σε μπουκάλια που θα πεταχτούν μετά, άρα λοιπόν και διανομή νερού και με ανθρακικό ας πούμε και αυτό μπορεί κανείς να το πάρει ένας πολίτης ακριβώς από τους κατάλληλους διανομής και να αποφύγει να αγοράζει εμφιαλωμένα νερά και άλλες παρόμοιες ενέργειες ώστε από το ξεκίνημα ήδη να μειώνουμε τα απορρίμματα και τα απόβλητα γενικά. Με το σχέδιο αυτό απαντάμε στις αναφορές που ήδη συζητήθηκαν στην πρόσφατη συνάντησή μας. Ποιο είναι το σημαντικό να γνωρίζετε ότι είχαμε διάφορες ενέργειες που επηρέασαν πραγματικά την κατάσταση από πλευράς τοπικής ε, αστυνομίας αλλά και νομαρχιακής αστυνομίας στην Ιταλία εκεί γίνεται ο συντονισμός των δυνάμεων της τάξεως ε, σε περιφερειακό επίπεδο, επαρχιακό επίπεδο και για όλες τις επαρχίες της Καμπανίας, κυρίως στην Νάπολη και στην Καζέρτα, όπου παρουσιάζεται ιδιαίτερα η εγκατάλειψη αποβλήτων και η καύση ανεξέλεκτη αυτών, εκεί υπήρξαν συμφωνίες ε, και μαζί με τις ε, καραμπινιέρους της περιοχής της ε, οικολογικής προσπάθειας και την δημοτική αστυνομία κατάλληλες συμφωνίες ακριβώς για να υπάρξει περισσότερη επαγρύπνηση όσον αφορά την, ε, τα, απόβλητα. Κάτι που ιδιαίτερα ελκύει την προσοχή και μάλιστα σε αρκετές αναφορές είναι η καύση μαζική αποβλήτων και πολλές φορές γίνεται και με ελαστικά αυτοκινήτων έτσι μαζικά πολλές φορές εμείς η Ιταλική κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος με ένα υπουργικό διάταγμα ε, όρισε ένα σύστημα ακριβώ όπως για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα δηλαδή υποχρεωτικά από το αρμόδιο εργαστήριο που πάνω από τον καράζ ακριβώ που αλλάζει τα ελαστικά σε ένα αυτοκίνητο ε, για να σου αλλάξουν τα ελαστικά σου πληρώνεις και ένα ποσό σου κρατάνε τα παλιά και με το ποσό που σου έχουν κρατήσει διαθέτουν έτσι τα καταστρέφουν τα ελαστικά όπως πρέπει και όχι μαζικά καύση ελαστικών που σημειωνόταν ε, άλλα χρόνια. Νομίζω ότι έτσι καλύψαμε σχεδόν τα πάντα όσα σας είπαμε. Απλευράς της κυρίας Ματσόνη αυτά που υπόθηκαν να τα επιβεβαιώσω γιατί είχαμε συμμετάσχει τις 15 Φεβρουαρίου με ε, Μαγκανάρο και Αλφιέρη είχαμε συναντηθεί και μάλιστα ε, ανταλλάξαμε και πάρα πολλές πληροφορίες και τις 15 Απριλίου με την προθεσμία αυτή, ακριβώς θα, στην προθεσμία αυτή μέσα θα στείλουμε μία έκθεση των νόσων των πεπραγμένων και το Υπουργείο Περιβάλλοντας ακριβώς θα ήθελε να τονίσει το πνεύμα διαφάνειας που μας χαρακτηρίζει αυτό θέλουμε να ισχύει στις σχέσεις μας και με τους πολίτες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια όχι μόνο στην περιφέρεια της Καμπανίας ε, με κέντρο την Νάπολη, αλλά παντού σε κάθε τοπική αρχή. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλετε να μου απευθύνετε κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα, ναι. Ναι, ναι, μετά, μετά η απάντηση. Σας ευχαριστούμε προς στιγμή όμως. Να προχωρήσουμε τώρα. Το λόγο έχει ο Δημοτικός Σύμβολος από το Μπενεβέντο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σε λίγα λεπτά μέσα θα προσπαθήσω να σας ε, πω με ποιους τρόπους εργαζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια. Δυστυχώς ε, πάντα ήταν ε, δύσκολη κατάσταση και παραμένει δύσκολη αλλά προσπαθούμε. Τώρα νομίζω ότι ερμηνεύω και τα όσα λένε και άλλοι και υπάρχει μια βεβαιότητα από πλευράς ρυθμιστικής και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πάνω σε ορισμένους χαραγμένους δρόμους ε, εδώ σχετικά με τον προγραμματισμό και τα πρώτα συγκεκριμένα που πετύχαμε σαν στόχους ε, Τώρα, μετά από μερικούς μήνες, δεν ξέρουμε εάν οι Ιταλικές επαρχίες τι θα γίνει, τι μορφή θα έχουν και ποια θα είναι η λειτουργία τους. Είναι κάτι που επηρεάζει την κατάσταση, ναι. Δυστυχώς χρειάζεται να το τονίσω για να σας πω πώς πέρα από ένα σταθερό προγραμματισμό Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι του να εμφανιστούν ρυθμιστικά πλαίσια τα οποία σε κανένα από εμά δεν επιτρέπουν δυστυχώς να πραγματοποιήσουμε τους στόχους πάνω στους οποίους εργαζόμαστε. Στον Πενεβέντο έχουμε περίπου 300.000 κατοίκους σε 78 δήμους. Και με τη διαφορμή συλλογή έχουμε μέχρι το 2010 είχαμε εκτός από το 42% τουλάχιστον το 2011 ε, θα πρέπει να το ελέγξουμε. Είναι σχεδόν βέβαια το στοιχείο αυτό. Είμαστε περίπου στο 55% αυτής της διαφοροποιημένης συλλογής. Το όριο που θέτει ο νόμος για το σύνολο της Ιταλίας. Άρα λοιπόν, για να υπάρχει μια σταθερότητα, πρέπει να ισχύει το ανώτατο όριο το 50%. Και είναι ιδιαίτερα πιθανό ότι το 65% το αποτέλεσμα που προβλέπεται για τις 31 Δεκάτου του 2012, ίσως, ίσως ε, το φτάσουμε αυτό, το 35%. Και ταυτόχρονα ε, μειώθηκαν όμως ε, στις χωματερές μας ε, τα φορτώματα εκεί αυτό το τελευταίο, αυτούς τους τελευταίους μήνες. Λοιπόν, Υπήρξε παρόλα αυτά διαμαρτυρία για, την, ε, για τον προγραμματισμό, αλλά προβλέπεται όμως εκεί η δυνατότητα να απομακρυνθεί κανείς από ένα κύκλο που είναι αποκλειστικά και μόνο επικεντρωμένος πρώτα απ' όλα στο άνοιγμα νέων χωματερών και ακόμα στο λειτουργία νέων αποτεφρωτών. και η δικιά μας πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη όσον αφορά τον πληθυσμό και με προσπάθειες ώστε το Μπενεβέντο να αποτελέσει ένα πρότυπο πολλές φορές ε, διαμαρτυρήθηκαν, αντέδρασαν όταν με συγκεκριμένα στοιχεία είπαμε ότι η μοναδική χαμετερή στο Σανταρκάντζελο Τρεμόντε θα έπρεπε να είναι κανονικά η τελευταία χωματερή στο Μπενεβέντο και μας το επιβεβαιώνουν αυτά οι αριθμοί. Αλλά ναι, και υπήρξε μια συντηρητική κατάσχεση από πλευράς ε, δικαστικών αρχών και ε, αυτό έγινε γιατί πήγε σε ένα μέρος που, υπήρχαν, που υπήρχε ένας γκρεμός και θα γκρεμιζόταν τα πάντα από κάτω. Α, λοιπόν, εδώ ε, δεν υπάρχει χωματερή πια στον Μπενεβέντο και αυτό δεν ε, δημιούργησε κανένα άσκημο καινούργιο παρόλο αυτό τον παραγωγικό κύκλο στον Πενεβέντο. Και ελπίζουμε ότι οι δικαστικές αρχές στις 28 ακριβώς αύριο θα μας ε, δικαιώσει στα όσα μέτρα λάβαμε. Παρά το ότι δεν έχουμε χρήματα, παρά τις δυσκολίες και τις διαθωτικές που αντιμετωπίζουμε, έγιναν πολλές εργασίες για την ασφάλεια και χάρη στην ε, ε, καλή διάθεση του διαχειριστή και επίσης ένας έλεγχος για το περιβάλλον και κυρίως όσον αφορά το νερό εκεί κοντά στη χωματερή και τα δείγματα έδειξαν θετικά αποτελέσματα μαζί και τον έλεγχο από τον σχετικό φορέα το Μάρσεκ μέσω δορυφόρου από τον Ιούλιο του 2011 μέχρι σήμερα ε, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες κινήσεις, αλλαγές. Εμείς περιμένουμε βέβαια με ελπίδα αλλά και αγωνία το αποτέλεσμα τι θα, κάνει, τι θα κάνουν οι δικαστικές αρχές, γιατί θα μπορούσαμε να βοηθάμε βοηθηθούμε και επίσης για μια οικονομική επίσης ε, σταθερότητα που διαφορετικά θα έπρεπε να επομισθούν οι αρχές του Μπενεβέντο και οι πολίτες. Λοιπόν, εδώ να σας πούμε ότι όλα αυτά τα κάναμε και τις τελευταίες εβδομάδες στην Καμπανία. Συναντηθήκαμε και με, την, με εκπρόσωπο της Ρώμης. Θα σας πω σχετικά μερικά πράγματα. Οι σχετικοί προγραμματισμοί κόστησαν πολύ λίγα χρήματα στην Πενεβέντο γιατί χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα που έχουν οι συνεταιρισμοί ακριβώς. Όταν ορισμένοι από εμά αγοράζουμε ε, ένα περίβλημα, ένα κουτί, κάτι τέλο πάντων και αντιμετωπίσαμε αρκετές δύσκολες καταστάσεις με 126 άτομα εργαζόμενους θα πρέπει να το επενθυμίσουμε αυτό γιατί στον προγραμματισμό μας εμείς ε, ε, καταφύγαμε, αλλά τελικά διακόψαμε, δεν ισχύουν πια δύο προκηρύξεις διαγωνισμών. Πρώτα απ' όλα για μια πλήρη υπηρεσία, θα ισχύουν για 10 χρόνια, με 212 εκατομμύρια ευρώ και για το τάσου για την αποκομιδή αποβλήτων. Ε, και όλα αυτά όμως βλέπουμε τα έχουμε και πάλι επειδή δεν υπάρχει μια αβεβαιότητα ρυθμιστική. Και εμείς είχαμε προβλέψει επίσης την ε, πλήρη απορρόφηση των 126 θέσεων εργασίας εργαζομένων που σε περίπτωση που θα έπρεπε να αλλάξουν τα πράγματα διαφορετικά δεν θα έβρισκαν καινούργια θέση εργασίας και βλέπουμε ότι θα λύνουμε πρόβλημα, θα ανοίγαμε ένα καινούριο. Και επίσης ε, Είδαμε τα διάφορα προβλήματα από τις οικολογικές ε, μπάλε, ας πούμε, ας τις αποκαλέσουμε έτσι, και για την εξυγίαση διαφόρων παλιών χωματερών που τα 15 χρόνια που προσπαθήσαμε να λύσουμε πηγόντως τα προβλήματά μας ε, λειτουργούσαν. Εδώ για να τις ε, ασφαλίσουμε αυτές τις χωματερές χρειαζόμαστε τουλάχιστον 17, να μπούμε και 19 εκατομμύρια που, ε, που δεν δόθηκαν όμως με υπουργικό διάταγμα αυτά τα χρήματα όταν λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις και ακόμα για να βρούμε αυτά τα χρήματα ας πούμε τι θα γίνει ε, δεν ξέρω ε, δεν θέλουμε να τα συμπεριλάβουμε στους φόρους που επιβάλλονται για να μην δυσκολέψουμε τη ζωή των φορολογουμένων. Εδώ. Προσπαθήσαμε από πλευράς να ενοποιήσουμε το πρόγραμμα ειδικών αποβλήτων με τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι ουσιώδες για μας θέμα, γιατί αυτά τα ειδικά απόβλητα αποτελούν τα δύο τρίτα της συνολικής ποσότητας, αλλά και του τι θετικού μπορεί να παραχθεί επί τόπου και τη στιγμή προωθούμε ένα σχέδιο μετά από μια Ιταλική συμφωνία μοναδικό στην Ιταλία με 15 φορείς που συμμετέχουν ε, τα κονσότσιουμ ακριβώς τα μεγαλύτερα με την ενοποίηση ειδικών αποβλήτων και αδρανών επίσης και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια αγορά μέσω του Green Public Procurement και επίσης ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας των αποβλήτων και προσπαθούμε έτσι να δούμε στο μελλοντικό σύστρι τι θα γίνει και πώς θα συμπεριφθούν. Θα την υποστηρίξουμε αυτή την ανιχνευσιμότητα με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα και το πρότυπο El του Σανίου και θα μπορούσε να συμπεριλάβει και άλλους χώρους να πάει και σε άλλες περιοχές. Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε. Ε, κάνουμε αυτά τα πειράματα, στα πούμε έτσι, και σημαντικό βήμα αποτελεί, και εδώ ολοκληρώνω, ολοκληρώνω, θα πρέπει να δούμε νέες εγκαταστάσεις που απαιτούνται για να πετύχουμε τους στόχους που ανέφερα προηγουμένως και για ένα διαφορετικό κύκλο αλλά να εναρμονίζεται με τον όλο περιφερειακό προγραμματισμό. Μέσω και του στήρου του Καζαλντούνη μια αλλαγή και είχαμε 56 εργαζόμενους εκεί, μεταφέρθηκαν και για το δικό μας παραγωγείο κύκλο κανονικά είχαμε ανάγκη από λιγότερους από τους μισούς αλλά εντάξει τους βρήκαμε νέα θέση εργασίας και σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τη συμπλήρωση μιας βιοσταθεροποίησης και έτσι θα βελτιώσουμε την ε, ποιότητα του παραχθέντος προϊόντος με λιγότερη ποσότητα αλλά στο Σαρκάζο Τριμόντε επειδή έκλεισε η χωματερία αυτή ε, βλέπουμε ότι φορτώθηκαν τελικά απόβλητα εκεί παραδίπλα και γι' αυτό ε, θέλουμε να επιτεχύνουμε την διαδικασία για να μπούμε στην τακτική διαδικασία. Και προφορικά με τον υπεύθυνο από το Δημοτικό Συμβουλίο της Ρώμης κλείσαμε μια συμφωνία και να δούμε την ε, ολοκληρωμένη αναεροβική εκμετάλλευση με συμπίκνωση του προϊόντος, πολτοποίηση και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε όχι μία τρομερά μεγάλη κατάσταση, αλλά διάφορες μικρότερες, γιατί και για τα ειδικά απόβλητα στη συμφωνία αυτή πρέπει να δούμε γεωργικές παραγωγές πώς συμμετέχουν και από τεχνικής πλευράς τι διαπιστώσαμε και χάρη στις ε, τεχνικές μας δυνατότητες ε, και της δρόμης επίσης, πώς θα μπορούμε όλα αυτά να τα προωθήσουμε. Και ένα ακόμα του Μολυνάρα, της Μολυνάρα που δεν λειτουργήσε ποτέ, πώς θα λειτουργήσει. Είχαμε 10 εκατομμύρια ευρώ για να ξεκινήσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις όπως ε, είχε καθορίσει καμπανία για τον Πενεβέντο και δυστυχώς δυστυχώς ζητήσαμε από τις τράπεζες να μας δώσουν χρήματα που θα μας εξυπηρετούσαν για να προχωρήσουμε αυτές τις κατάσταση. Αλλά καμία τράπεζα παρά τις εγγύησεις και παρά το ότι έτσι κι αλλιώς αυτοτροφοδοτούνται αυτά τα ποσά σε δεύτερη φάση. Καμία τράπεζα δεν δέχτηκε να συμμετάσχει σε αυτές τις επενδύσεις και θέλω να το τονίσω. Τις εβδομάδες που ακολουθούν ε, και εμείς θα ξεκινήσουμε με μια, ένα πρόγραμμα μείωσης των αποβλήτων. Στον Πενεβέντο είχαν αφιερώσει ήδη 50.000 ευρώ και αυτά που είπε ο, Σαν, Σαντακρότσε πριν από μένα και χάρη στην ε, βοήθεια της περιφέρειας ε, της Καμπανίας θα διπλασιάσουμε το ποσό αυτό και να δούμε πώς ε, θα μπορούσε να υπάρξει ένα σύστημα αποβλήτων που να περνάει μέσω από τη μείωση των αποβλήτων και να μπορούμε να έχουμε και μια ανακύκλωση και να δούμε και... Εντάξει, έχουμε, διαθέτουμε ένα πρόγραμμα και τις ε, επαρχίας και το βιομηχανικό. Και βλέπουμε από τεχνικής πλευράς τι μπορεί να γίνει με αυτά τα προγράμματα και νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να προχωράμε, τα ταυτόχρονα να είμαστε και αποφασισμένοι για να δούμε και καινοτόμες εγκαταστάσεις αποδοτικές. Ευχαριστώ. Γκαμπακόρτα από Αβελίνο, Δημοτικός Σύμβουλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε για τη δυνατότητα την οποία μας προσφέρετε γιατί κάνουμε ένα υπολογισμό ακριβώς της δραστηριότητας του Αβελίνο σε συμφωνία με την περιφέρεια της Καμπανίας και συνεργασία με άλλες επαρχίες της Καμπανίας το 2010, το 2011 που είναι ακριβώς οι δύο χρονιές μας απασχόλησαν ιδιαίτερα μετά από τη μακρά περίοδο κρίσης και της μεγάλης ποσότητας αποβλήτων στην περιφέρεια της Καμπανίας. Είδαμε τις αναφορές, ορισμένες από αυτές ε, έχουν να κάνουν με την περιοχή του Αβελίνου. Θα μιλήσω για αυτές. Και εμείς είχαμε την, ε, προχωρήσαμε στη σύσταση του Φορέα για την προστασία των πολιτών από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και ακριβώς ε, είναι υπεύθυνος ο Φορέας αυτός και για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων στην περιοχή μας όπως επίσης και για την υπηρεσία διαφοροποιημένης συλλογής των αστικών αποβλήτων σχεδόν σε όλη την περιφέρεια του Αβελίνο, το 85% των δήμων εκεί. Θα πρέπει να τονίσουμε κάποια αποτελέσματα που αυτά τα χρόνια πετύχαμε. Πρώτα απ' όλα η διαφοροποιημένη αυτή συλλογή, τα στοιχεία που είναι ιδιαίτερα ενδεικτικά. Στην περιφέρεια του Αβελίνο είχαμε φτάσει ήδη το 48,78% διαφοροποίηση συλλογή το 2009. Και αυτό έχει να κάνει και με πολλούς μικρούς, πολύ μικρούς δήμους της ε, επαρχίας μας, αλλά και στην τοπική πρωτεύουσα είχαμε ένα υψηλό ποσοστό. Το 2010 το ποσοστό αυτό ε, αυξήθηκε, πήγε στο 51,23% και χαρή και στην ε, βοήθεια της πρωτεύουσα που έφτασε στο 62 και κάτι της 100, Βέβαια δεν είναι επίσημη ακόμα η αριθμή, αλλά ξεπεράσαμε και πάλι το 5% μιας διαφοροποιημένης συλλογής και 79 από τους Δήμους που είναι διπλάσιοι έφτασαν το αυτό που αναφέρεται από το νόμο 123 αυτό το 50 και κάτι και αρκετοί δήμοι πήγαν και στο 70% και ακριβώς ο φορέας της ε, περιοχής του Αβελίνο σε όλους σχεδόν τους δήμους για το 2012 θα, μπορούσε, θα μπορέσει να συλλέξει τα απόβλητα μέσω ενό συστήματος από έτσι μέτρο μέτρο να το κάνει προχωρώντας ε, με επίσης δίδονται πριν ε, για όσους πετυχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα αλλά επίσης και κύρος εφαρμόζομαι για τους Δήμους που δεν έφτασαν τις ε, νόμιμες προβλέψεις γιατί όσον αφορά την επεξεργασία των αποβλήτων ε, που δεν το έχουν πετύχει αυτό, απαιτείται υψηλότερο κόστος. Και επίσης το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε για τις χωματερές. Υπάρχουν τρεις χωματερές στο Αβελίνο. Ένα μια χωματερή που σχεδόν έχει κλείσει και άλλες δύο που υπάρχουν ακόμα. Σχετικά με την αμπρέτα, τη χωματερή αυτή, αυτή να αναφέρει μια αναφορά ακριβώς προβλέπεται από το ε, διάταγμα του 90 και ανανεώθηκε το 2008. Με το 2011 νόμο 1 βλέπουμε ότι ε, δεν προβλέπεται πια στην περιοχή Φορμικόσο η χωματερή και ακόμα μια χωματερή για την οποία διαμαρτύρονται οι αναφέροντες ήταν στην Τιφέζα Γκράντε από το 2007 όμως έχει κλείσει κανονικά επιχειρησιακά, αλλά και χάρη σε ένα νόμο την 5η Ιουλίου του 2007, την 87 νόμο, που έκλεισε έτσι οριστικά αυτή η χωματερή. Το 2011 είχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ε, σε αυτές τις ε, ε, ανάμεσα στους δύο. Η χρηματοδότησε για την βελτίωση όλων αυτών με 6,5 εκατομμύρια ευρώ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος τώρα ζήτησε από την ε, περιφέρεια αυτή βάσει του άρθρου 244 του 155 νομοθετικού διατάγματος να ρυθμιστούν τα πράγματα. Επίσης έχουμε την ε, χωματερή του Σαβινιάνο που εξυπηρετούσε το 2008 και 2009 το σύστημα αλλά έχουμε μια τρομερή μείωση πραγματικά αποβλήτων από 50.000 τόνους το μήνα το 2008 περάσαμε στους 30.000 τόνους το 2009 και 10.000 ε, τόνους ακόμα το 2011 το 2010. Το 2011 είχαν ε, όλες και όλες 68.000 τόνους όλο το χρόνο και εμείς ε, προσέχουμε ιδιαίτερα τις ανάγκες της περιοχής και είχαμε μια διαχείριση στο Αβελίνο και χάρη στην διαφοροποιημένη αυτή συλλογή αλλά έτσι ακριβώς μπορούμε να σεβαστούμε και την επαρχιακή αυτάρκεια, όπως επίσης να σεβαστούμε και την αρχή του πώς θα είναι κοντά αυτοί που ξεφορτώνουν αυτά τα απόβλητα και όχι να έρχονται από μακριά γιατί από μακριά μεταφορές αποβλήτων δημιούργησαν τρομερές δυσκολίες και προβλήματα. 2010-2011 είχαμε μια διαχείριση όπως είπαμε από ένα δημόσιο φορέα και καθυσίχασε έτσι τους πολίτες και μαζί με το Σαβινιάνο, την τοπική αρχή ε, υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο συμφωνίας ε, ώστε να μειωθούν ακόμα περισσότερο τα απόβλητα εκεί στην ε, χωματερία αυτή. Κάτι που θέλω να τονίσω επιπλέον είναι ότι όταν η επαρχία έγινε ακριβώ η υπεύθυνη, η αρμόδια και υπεύθυνη για τον κύκλο αυτό αποβλήτων στην περιοχή μας, 14.000 Μπάλε, α πούμε έτσι είχαμε κληρονομήσει εισαγωγικά 25.000 τόνους περίπου και μειώσαμε τον όγκο αυτό κατά 10.000 και ένα σημαντικό μέρος πήγε για επεξεργασία οριστική στι ε, εγκαταστάσεις που παράγουν ε, θερμική ενέργεια. Και ακόμα ένα σημαντικό αποτέλεσμα το οποίο πετύχαμε το 2011, δύο εγκαταστάσεις εκεί στην επαρχία, είχαμε μέσω κατάλληλης διαδικασίας ε, συνήθως διαδικασίες ε, να προχωρήσει και θα έχουμε στη Μοντέλα να δούμε την διαφοροποιημένη συλλογή ξηρών αποβλήτων 22 Δεκεμβρίου του 2011 απόφαση. Το ίδιο ισχύει και για το πιάνο Ντάρντινε που τις 5 Δεκεμβρίου του 2011 με διάταγμα ακριβώ πήρε την ε, άδεια για παρόμοια διαδικασία για να να αποτελέσει κέντρο αναεροβικής επεξεργασίας όσων παράγονται στο Αβελίνο για περίπου 30.000 τόνους το χρόνο. Και βέβαια, ολοκληρώνοντας τώρα, μετά από τη δημοσίευση του περιφερειακού σχεδίου με τον περιφερειακό προγραμματισμό, ήδη υιοθετήσαμε το σχετικό έγγραφο του Σκόπιν για το περιφερειακό πρόγραμμα αστικών αποβλήτων και είμαστε έτοιμοι να δημοσιεύσουμε την σχετική έκθεση μετά από την στρατηγική ανάλυση από την ε, πανεπιστήμιο που έχει συνταχθεί της περιοχής ε, και στο Αβελίνο στο σύστημα πέρασαν 7 εκατομμύρια ευρώ ήδη πόροι για να αντιμετωπιστεί το κόστος στον τομέα αυτό γιατί κοστίζει χρήματα η διαφοροποιημένη συλλογή και η φορέας για το περιβάλλον χρειάζεται πολλά χρήματα σε μια βάση. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν ότι εργαζόμαστε ιδιαίτερα έντονα για να εγγυηθούμε και μια αλληλεγγύη και σε άλλες περιοχές όπως το 2010 και το πρώτο μέρος του 2011 υπάρχουν ανάγκες οικονομικές για να ανέβουμε τα αποτελέσματά μας και δυστυχώς επειδή ξέρουμε πως έχει όλη η διαδικασία παράβασης έχουν παγώσει οι σχετικές πιστώσεις και μιλήσαμε για τις παλέτες που έχουμε εκεί στις χωματερές δίπλα αυτά τακτοποιούνται και για το βιομηχανικό πρόγραμμα του φορέα αυτό τίθεται ο στόχος του 65% για το 2012, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από το κασονέτο μέχρι το, αυτό το βήμα-βήμα που κάνουμε, όλα αυτά πράγματα μας δείχνουν ότι έχουμε 75% περίπου και πάνω συλλογή. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, και τώρα το λόγο έχει ο Δημοτικός Σύμβουλος Φορτουνάτο από την επαρχία του Σαλέρνου. Καλησπέρα. Θα ήθελα να χαιρετήσω και εσάς κυρία Πρόεδρε από πλευράς του Δημόντο Σιβίλ, ε, του Πρόεδρου που δυστυχώς αδυνατεί απόψε να παραστεί και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω όλους και το σύνολο της Επιτροπής περιβάλ ε, συγγνώμη, Αναφορών. Να περάσω στο κύριο θέμα για το πώς έχουν τα πράγματα στο Σαλέρνο. Στην Καμπανία είναι ο δεύτερος δήμος, δήμος 2.200.000 κάτοικοι, 158 δήμοι. Αλλά είμαστε και οι καλύτεροι όσον αφορά τη με συλλογή. Το 2010 είμαστε περίπου στο 55%. Το 2011 πήγαμε κάνοντας και τους λογαριασμούς μας, τους υπολογισμούς μας, ε, θα φτάσουμε στο 65% τώρα. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Ότι στην περιφέρεια της Καμπανίας υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, αλλά υπάρχουν και πολύ καλά σημεία. Άρα λοιπόν, αν δούμε το σύνολο μιας περιοχής θα πρέπει εκεί να λέμε και τα πράγματα που πάνε χάλια, εντάξει να το πούμε, να το αντιμετωπίσουμε, αλλά και πράγματα που πάνε πολύ καλά όπως στη δικιά μου περιοχή, στην περιοχή του Σαλέρνο. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το συντάκτη της ε, αναφοράς ε, ο κύριος Βιντσέντζο Μάρμορα, γιατί εδώ είμαστε για να απαντήσουμε σε αυτή την αναφορά και για την επαρχία του Σαλέρνου για την 27 του 2007 από τον κύριο από την κυρία Μόνικα Σέπε για ένα σχέδιο μιας ε, ε χωματερής στη Βάλεντε Λεμασερία. Μπορώ να σας πούμε με ιδιαίτερη μας χαρά και ικανοποίηση βέβαια ότι η επαρχία του Σαλέρνο ανέλαβε την υποχρέωση και το έκανε και μπροστά στην Επιτροπή που έκανε τους σχετικούς ελέγχους ε, για να κλείσουμε στη Βάλντελα Μασερία τη χωματερή αυτή και με το 196 του 2010 με το σχετικό νόμο, άρθρο 1, εδάφιο 1, ε, με το διάταγμα αυτό κλείνει αυτή η χωματερή Θέλαμε να το κάνουμε, είναι πραγματικά ιδιαίτερη σημασία αυτή η χωματερή για μας, αρνητική σημασία. Λοιπόν, για τον Μπάσο Ντελόλμο, αυτή έχει γεμίσει. Έχουμε ένα έλεγχο μέσω του περιφερειακού φορέα και προσέχουμε ιδιαίτερα τι γίνεται εκεί για να σεβαστούμε τη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν για την επαρχία του Σαλέρνου αυτά, όπως επίσης και στη Λαμασερία στην χωματερία αυτή που είπαμε όχι, Μάκια Προβάνα. Και έχουμε μια διαχείριση από το κονσόρτσιουμ το αρμόδιό είναι αρμοδιότητα της επαρχίας του Σαλέρνου άρα λοιπόν για αυτή τη χωματέρη για τις χωματερές μπορούμε να σας πούμε ότι τις ελέγχουμε όλες, προσέχουμε ιδιαίτερα και το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Ακόμα κάτι το σημαντικό είναι, θα πρέπει να το πούμε και θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλη την Επιτροπή σας και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η περιφέρεια της καμπανίας, γιατί είμαι και σύμβουλος της περιφέρειας, εγκρίναμε στο Συμβούλιο αυτό το πρόγραμμα το οποίο υπήρχε η απέτηση να εγκριθεί, τελικά το κάναμε και θα πρέπει να τονίσουμε το ότι εμείς οι καθημερινοί πολίτες αλλάξαμε την ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον και όπως στο Αβελίνο Μπενεβέντο ε, και στο Σαλέρνο βλέπουμε ότι ε, κάναμε τον κόσμο να έχει μια διαφορετική εικόνα και αντίληψη σχετικά με τα απόβλητα και να καταλάβουν όλοι ότι χρειάζεται μια κοινή προσπάθεια πάνω απ' όλα για την εξειδικευμένη συλλογή. Και εμείς όλοι το κάναμε αυτό, μέτρο-μέτρο μπορούμε, πηγαίνουμε, μπορώ να σας πω. Και πριν μερικού μήνες ακόμα ήμουν δήμαρχος. Ακόμα και τα τζάμια τα σπασμένα πάμε και τα παίρνουμε. Και φτάσαμε και μέχρι το 85%. Υπάρχουν ε, πραγματικά ιδιαίτερα προχωρημένοι δήμαρχοι Εμεί στο Σαλέρνο, 85% και εμείς όμως ξεκινήσαμε ε, σε μερικά μέρη και πιο αργά, αλλά και εκεί τα κατάφεραν. Για το μέλλον ε, τρέφω την πίστη ότι αυτό αποτελεί ένα καλό μάθημα. Ναι. Εδώ ίσως είναι πιο ρότερη περιοχή της Ιταλίας στην Καμπανία και στη Μεσόγειο αλλά με την κακή διαχείριση στο παρελθόν έχουμε χαλάσει πάρα πολύ την εικόνα μας επειδή έχουμε μια νέα ε, νέες αρχές προωθούμε, προχωράμε, βοηθάμε. Και για να αλλάξει αυτή η εικόνα, εντάξει, είμαι πεπισμένος ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα και βέβαια με ατενίζοντας ε, και προσέχοντας και αυτά που μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας καθοδηγεί θα μπορούσαμε να πετύχουμε το στόχο μας και να βγούμε αυτή την τρομερά σκημη κατάσταση που κατέστρεψε όσους δεν μπόρεσαν να τα διαχειριστούν αλλά και ακόμα και καλές περιοχές τους έκανε ζημιά στην εικόνα τους όπως στην περιοχή του Σαλέρνο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν ε, ο συνάδελφος ε, μηχανικός Ντακούντσι θα συνεχίσει αλλά όσον αφορά την επαρχία του Σαλέρνο θα είμαστε εντελώς ε, αυτόνομοι σε δύο-τρία χρόνια γιατί και στην πόλη του Σαλέρνο έχουμε μια θερμική επεξεργασία και σαν περιφερειακό σύμβολος να σας πω ότι είχε αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου. Υπάρχει διάθεση να πετύχουμε αυτό το ποιοτικό άλμα για νέα αξιοπρέπεια στην Ιταλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς είμαστε μέλη αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Εδώ οι προηγούμενες παρεμβάσεις ακριβώς σίγουρα θα σας έκανα να καταλάβετε ότι είμαστε στη φάση της εφαρμογής του προγράμματος. Αυτό το πρόγραμμα για τα πόβλητα και εγκρίθηκε αλλά εφαρμόζεται και μπορέσαμε μάλιστα να τρέξουμε και γρηγορότερα από ό,τι είχε προβλεφτεί γιατί υπήρχαν ήδη τα βιομηχανικά σχέδια που με ρύθμιση κατάλληλη σε επαρχιακό επίπεδο και φορείς που προχωρήσαμε στη σύστασή τους ακριβώς αυτές τις δύσκολες στιγμές για τον ολοκληρωμένο κύκλο. Εδώ που παίζεται το παιχνίδι στην γοργή πραγματοποίηση, εγκατάσταση όλων αυτών που να έχουν όμως αποτέλεσμα να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνολογία αλλά και πάνω απ' όλα τη δυνατότητα να ικανοποιήσει κανείς τον ε, κύκλο αυτό και ο πληθυσμός ε, που είναι εκεί κοντά να μπορεί να κάνει το σχετικό έλεγχο, πραγματικό, αντικειμενικό, πώς γίνεται η όλη διαχείριση και λειτουργία. Σχετικά με την επαρχία του Σαλέρνου αυτή η διαφοροποιημένη συλλογή είναι στο ύψος του 54-55% του μεσουόρου που είναι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Για το 11 και 12 περιμένουμε ακόμα υψηλότερα ποσοστά. Για να είμαστε στα 158 δήμους, μόνο 16 δήμοι δεν έχουν φτάσει στο 35%. Ξέρω αυτό για να είμαστε και ακριβείς. Έτσι, 158 ναι, 13, στο σύνολο 158, 13 όχι. Και προωθούμε μία άμεση παρέμβαση και με υπαλλήλους μας που πηγαίνουν επί τόπου βλέπουν που είναι το δύσκολο σημείο και βοηθούν για την ε, χάραξη προγραμμάτων ε, για να βοηθήσουν και εμείς ε, διεξάγουμε μελέτες για να έχουμε μια συλλογή ποιοτική επίσης και από τη στιγμή που φτάνουμε σε αυτό το ποσοστό, το καινούριο πρόβλημα ποιο είναι. Αυτές τις ποσότητες, αυτά τα απόβλητα που παίρνουμε, να τα αλλάξουμε και τα κάνουμε πρώτη ύλη. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε την σχετική τεχνολογία ώστε να προχωρήσουμε σε ιδιωτικές και δημόσιες παρεμβάσεις για να εκμεταλλευτούμε τα απόβλητα αυτά που έτσι μεικτά συλλέγονται. Αυτό και για το οργανικό μέρος των αποβλήτων που είναι από τα μεγαλύτερα μας προβλήματα. Είδαμε ότι 113.000 το χρόνο απόβλητα οργανικά χρειαζόμαστε να... Ε, ε, ε, και έχουμε ένα σύνολο 140.000 τόνων και έχουμε πέντε εγκαταστάσεις ε, που θα πρέπει να αναπτυχθούν για να αποφύγουμε και τη μεταφορά αυτών των οργανικών αποβλήτων από μία περιοχή στην άλλη. Μία εγκατάσταση ολοκληρώθηκε στην ίδια την πόλη του Σαλέρνο. 30.000 τόνοι η επεξεργασία το χρόνο. Το εργοστάσιο αυτό έχει προχωρήσει, έχει ξεκινήσει και θα δεχτεί πολύ ψηλέ ποσότητες ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες ε, του συνόλου της πόλεως και της περιφέρειας του Σαλέρνο. Επίσης άλλη μια εγκατάσταση εκεί κοντά στο Έμπολι, στο Έμπολι είναι για 20.000 τόνους ε, στην πόλη του έμπολι. το έμπολι. εκεί που σταμάτησε και ο Ιησούς, το έμπολι. Λοιπόν, εδώ να σας πω ότι υπήρξε μια προκήρυξη διαγωνισμού και το πήραν εταιρείε που θα προχωρήσουν στην κατάσταση αυτή τους επόμενους μήνες και ε, μόνο 30.000 τόνοι δεν καλύπτονται και έχει προβλεφθεί η σχετική επεξεργασία στο νότια πλευρά στο Βάλεντε Λαλουκάνια Εκεί θα τα επεξεργαστούν και εκεί θα έχουμε την πέμπτη, το πέμπτο εργοστάσιο 30.000 τόνων δυναμικότητας. Έχει ξεκινήσει το σχέδιο για να προκηρυχθεί και ο σχετικός διαγωνισμός που θα προκηρυχθεί ακριβώς τις μέρες που ακολουθούν. Αυτά για τα οργανικά απόβλητα για τη θερμική επεξεργασία που προβλέπεται στο Σαλέρνο τι θα πρέπει να πούμε. Αυτούς τους τελευταίους μήνες ε, της χρονιάς μας πέρασε, πολύ καλά προχώρησε η Επιτροπή για να αναθέσει οριστικά το εργοστάσιο έγινε τον Ιούλιο του 2011. Και ένας διαγωνισμός που δεν έχει προκηρυχθεί έχει να κάνει Πρώτα απ' όλα με ένα πιστοποιητικό αντιδιαφθοράς από τη δικαστική αρχή του Μιλάνου. Για τη θερμική επεξεργασία χρειάζονται τρία χρόνια για την εγκατάσταση. Τρία χρόνια εργασιών τα τρία χρόνια αυτά τι προβλέψαμε. Να ξεπεράσουμε την προπασκευαστική βάση, τη μεταβατική βάση και να έχουμε και περαιτέρω εγκαταστάσεις για μια καλύτερη διαφοροποιημένη συλλογή αλλά και την, πραγματο... και την εγκατάσταση τεσσάρων ε, χωματερών όμως ειδικών ε, για να πάρουν ε, τα απόβλητα από περιφερειακά και η επαρχία του Σαλέρνο χωρίστηκε σε τέσσερις τομείς που αντιστοιχούν λίγο πολύ στους δήμους των προηγούμενων οργανισμών φορέων για την επεξεργασία και θα μπορούμε να έχουμε έτσι τέσσερις μικρές χωματερές που για τρία χρόνια ακόμα θα μας επιτρέψουν να έχουμε εκεί τα απόβλητα αλλά τρία χρόνια δεν θα είναι κάτι που θα υφίσταται μικροβιακή ε, επεξεργασία παντού προσπαθούμε να έχουμε ένα βιοσταθεροποιητή για να έχουμε ένα απόβλητο που θα μας δίνει ένα συμπυκνωμένο σύνολο συγκεκριμένο και ε, ουσιαστικά αν υπάρξει διήθηση δεν θα είναι πλήρης. Αυτά λοιπόν και όλα αυτά για το καλό του πληθυσμού. Και για τις χωματερές να σας πούμε. Ναι, ναι, ολοκληρώνω με το νόμο 1 του 2011 ήδη έχει οριστεί ένας επίτροπος ο οποίος και θα πρέπει να δει και να ελέγχει αυτές τις χωματερές τις προσωρινές. Για αυτές τις τέσσερες χωματερές που βρήκε ο επίτροπος που διόρισε ο πρόεδρος της Περιφέρειας Καμπανίας έχουμε τα οριστικά σχέδια και θα προχωρήσουμε γρήγορα γρήγορα στην προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών. Έτσι κλείνει αυτός ο κύκλος με τα απόβλητα και μπορούμε να διαχειριστούμε ε, πλήρως ε, όλο τον κύκλο. Σας ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος, η πρόεδρος. Θα πρέπει να επιταχύνουμε όμως, ε, γιατί ξεφεύγουμε από το πρόγραμμα. Από την Άπολη Ναπολετάνο. Καλησπέρα σας. Πώς έχει κατάσταση στην επαρχία της Νάπολης. Εκεί κάπως χειρότερη βέβαια σε σχέση με τις υπόλοιπες. Επειδή υπάρχει και υψηλότερος πληθυσμός, αλλά υπάρχουν και διάφορα προβλήματα τυπικά της περιοχής. Γνωρίζετε ότι στην Νάπολη δεν έχουμε εγκαταστάσει επεξεργασίας ε, εκτός από τις τρεις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ε, με ένα μέρος ε, στεγνό ξηρό ε, τελικό προϊόν και ένα σχετικά υγρό. Και βέβαια για τη μεταφορά δεν υπάρχει ιδιαίτερη δυνατότητα γιατί και το ξηρό απόβλητα προέρχεται από τα Στυρ και από άλλες περιοχές Καμπανίας. Γιατί το Καγιάνο και στο Τερσίνιο, τις δύο χωματέρες ε, ε δυστυχώς έχουν σχεδόν γεμίσει προπαντός του Καγιάνο ε, έκλεισε μόλις ε, για διάφορες διαφθορτικές αλλαγές ενώ στο Τερτσίνιο οι χωματεροί αυτοί ε, φτάνουν φτάνει ακόμα η χωρητικότητα για δύο-τρεις μήνες το πολύ και πάει και αυτή γέμισε και στην Άπολη θα μπορούσαμε να έχουμε για τον όλο προγραμματισμό για αυτόν τον κύκλο αυτό αποβλήτων κατάλληλα ε, προγράμματα. Έστω και αν υπάρχουν ε, διάφορε ε, διάφορες δυσκολίες και άγνωστοι παράγοντες όπως είπε και ένα προηγούμενο ομιλητή, και υπάρχουν και δυσκολίε και έτσι η Περιφερειακή Αρχή δεν μπόρεσε να κάνει την κατάλληλο προγραμματισμό τουλάχιστον σε διετή ή τρίτη βάση αλλά στην επαρχία της Νάπολης Εκεί ενεργοποιηθήκαμε ιδιαίτερα και από το δικά μας χρήματα δώσαμε τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ τα τρία τελευταία χρόνια και για καλύτερες οικολογικές νήσους και για κατάλληλα μέσα μεταφοράς κλπ. Και είχαμε 64 οικολογικές νήσους και θα προβλέπονται κι άλλες. Έτσι να πραγματοποιήσουμε, να προχωρήσουμε το περιφερειακό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων. Επίσης ξεκινήσαμε με διάφορες τοπικούς φορείς, πρωτοβουλίες για να πετύχουμε το βασικό στόχο για αυτό ένα σύντομο κύκλο αποβλήτων, για να ανοίγει και να κλείνει ο κύκλος εκεί επιτόπου σχεδόν κάτι που μέχρι τώρα δεν το πετυχαίναμε. Και επίσης ε, χωρίστηκε σε 7 τομείς ομοιόμορφες ε, η περιοχή και είχαμε συμφωνίες μια προγράμματα και μακροπρόθεσμα θα έχουμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ώστε αυτοί οι τομείς ε, να είναι εντελώ αυτόνομοι στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων. Και στις περιοχές αυτές ε, μπορούν να υπάρξουν και χωματερές όχι για αυτά καθ' αυτά τα απόβλητα, α πούμε, αλλά στα στήρ να έχουμε βιοσταθεροποιητές που θα έχουμε βάσει και του κατάλληλου κώδικα. Ένα ε, πολτοποιημένο απόβλητο και κάπως συμπυκνωμένο και έτσι να δούμε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μάλιστα όσον αφορά τη μορφή τους και να έχουμε αυτό το βιοσταθεροποιημένο από τα στήρ της εγκαταστάσεις αυτές απόβλητα και θα τα καταφέρουμε από τα στήρα αυτά, από τις εγκαταστάσεις αυτές και το περιφερειακό πρόγραμμα τι προβλέπει την εγκατάσταση δύο αναεροβικών ε, εγκαταστάσεων. Σε κάθε, μία από αυτές, σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς θα έχουμε ένα-δύο εγκαταστάσεις ε, για πολτοποίηση και συμπίκνωση των αποβλήπων των και στα δύο χρόνια τα οργανικά απόβλητα θα μειωθούν πολύ και σε τρία χρόνια θα έχουν εξαφανιστεί. Και ακόμα στη διαφορεμένη συλλογή στην Νάπολη, βέβαια τα στοιχεία δεν είναι τόσο καλά όπως και στις υπόλοιπες περιφέρειες, ε, 2010 27% μόνο ε, Δυστυχώ, η ουσία των Δήμων δεν πέτυχε το 35% που είχε προβλέψει ο νόμο, πάντως και στην Άπολη είχαμε διάφορα πολύ θετικά αποτελέσματα που πέτυχαν αυτό το 35% αλλά και πολύ παραπάνω, 60-70%, 45% 60%. Βέβαια πίσω-πίσω δυστυχώς είναι η ίδια η Νάπολη που προσπαθεί, προσπαθεί όμως ώστε και μέσα στην πόλη της Νάπολης να έχουμε καλύτερη, περισσότερη διαφοροποιημένη συλλογή. Νομίζω ότι κάλυψα τα πάντα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρος. Φάλκεμπεργκ, από την Επιτροπή. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα. Εδώ και πολύ καιρό. Είναι μία από τις ε, χειρότερες ε, καταστάσεις ό,τι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων που, με την οποία ήρθαμε αντιμέτωποι. Αναγνωρίζουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, υπάρχει βελτίωση και χαιρόμαστε που η Περιφέρεια επιτέλους υιοθέτησε φέτος τον Ιανουάριο ένα ε, σχέδιο διαχείρισης ε, δημοτικών αποβλήτων ή αστικών αποβλήτων. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι αυτό έγινε πάνω από 1,5 χρόνο μετά την απόφαση του δικαστηρίου ότι η Ιταλία εφάρμοσε πλημελώς ε, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε αυτή την περίπτωση. Εξακολουθούν να υπάρχουν ε, ζητήματα που μας ανησυχούν και αυτό το ξεκαθαρίσαμε και στις ε, πρόσφατες επαφές μας με την Ιταλική κυβέρνηση. Ο Επίτροπος Ποτότσνικ συναντήθηκε με τον Υπουργοτενή τον Ιανουάριο. Και ποιες είναι αυτές οι ανησυχίες. Αυτές αφορούν το γεγονός ότι εξακολουθούμε να βλέπουμε στην περιφέρεια αυτή πολύ, μικρή, πολύ μικρό βαθμό διαχωρισμού των αποβλήτων, κάτι που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα σε αυτή την ε, περιφέρεια, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων. Ακούσαμε πολλά για την αναερόβια κομποστοποίηση πάνω από ένα χρόνο μετά την απόφαση μόνο μία επιπλέον ομάδα λειτουργεί και, τα, και οι υπόλοιπε μονάδες θα αρχίσουν να λειτουργούν ε, κάποια στιγμή από τώρα μέχρι το, την άνοιξη του 2014. Ε, υπάρχουν αποτεφρωτές που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν ε, το 2014 και το 2015. Επιπλέον ε, χώροι υγειονομικής ταφής δεν γνωρίζουμε κάτι από αυτού προς το παρόν και έχουμε και πάλι 7 εκατομμύρια τόνους εκομπάλε. Ε, την πολύ αυτή γνωστή κατηγορία αποβλήτων. Εμείς δεν είχαμε άλλη επιλογή. Πέρσι, στα τέλη του χρόνου, στείλαμε ακόμα μία ε, ε αποστολή προειδοποίηση αν θέλετε, προ την ε, Ιταλική κυβέρνηση. Βρισκόμαστε συνεχώ σε επαφή με την Ιταλική κυβέρνηση. Ε, στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να δούμε και να αξιολογήσουμε μήπως πρέπει να επιστρέψουμε στα δικαστήρια. Ιδίως γιατί βλέπουμε ότι έχουμε ανεπαρκή ε, μεσοπρόθεσμα μέτρα για, την, ε, για το σχέδιο διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Ακούσαμε και σήμερα ότι πολλές από τις εγκαταστάσεις αρχίζουν αρχίσουν να λειτουργούν κάποια στιγμή στο μέλλον και εντωμεταξύ χρειαζόμαστε ε, επαρκή μέτρα μέχρι τότε. το Περιφερειακό Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο για τα αστικά ε, απόβλητα, αλλά ακόμα περιμένουμε την έγκριση του σχεδίου για τα ειδικά απόβλητα. Εάν όλα αυτά δεν γίνουν μέσα στο πολύ πολύ άμεσο μέλλον, η Επιτροπή, όπως είπα, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει το επόμενο λογικό βήμα, δηλαδή να παραπέμψει και πάλι την Ιταλία στα δικαστήρια. Όμως ε, συνομιλούμε με την Ιταλική κυβέρνηση και θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε αυτή την κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Παρακαλώ συνάδελφοι όσοι έχετε εγγραφεί. Έχουμε πολλές εγγραφές εδώ. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Έχουμε καθυστερήσει πέντε λεπτά και από όσων είχε προβλεφθεί. Παρακαλώ, γρήγορα, γρήγορα. Χέλμερ. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των τοπικών ε, αρχών ε, από την περιφέρεια της Καμπάνια για την ε, πολύ καλή γενική εικόνα που μας έδωσαν για την κατάσταση αυτή. Δεδομένε τη διαδικασία υπεπαραβάση που κίνησε η Επιτροπή πριν από πέντε χρόνια, δηλαδή το 2007, με εκπλήσει το γεγονός ότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιος είναι ο αριθμός των εγκαταστάσεων, αλλά είναι σαφές ότι δεν είναι αρκετές και μόλις πρόσφατα εκπονήθηκε ένα σχέδιο και δεν υπάρχει περαιτέρω πρόοδος. Χαίρομαι που γίνεται όλη αυτή η αναφορά με, τη, με τους αποτεφρωτές και την ε, ανάκτηση της ενέργειας. Καλό αυτό αλλά αυτό μας οδηγεί και στο ζήτημα της ικανότητας. Ε, ακούσαμε πολλά μεγάλα νούμερα, αλλά και πάλι δεν έχω καταλάβει ποια είναι, η συνολική ικανότητα, capacity που υπάρχει και αν καλύπτει την ε, ζήτηση για την διάθεση αποβλήτων. Πολύ είδαμε και στις τηλεοράσεις μας πριν από, ε, πριν από μερικά χρόνια τις ορούς ε, σκουπιδιών ε, που συσσωρεύονταν στους δρόμους της ε, Νότιας Ιταλίας και θυμόμαστε και τον κύριο Μπερλουσκόνη που έκανε επισκέψεις και δηλώσεις επιτόπου. Θα ήθελα να ξέρω αν εξακολουθούν να υπάρχουν σωροί σκουπιδιών στους δρόμους ή αν τουλάχιστον έχει επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Ακούσαμε και για συμφωνίες με Ολλανδούς παρόχους υπηρεσιών στην ε, αποκομιδή και στη διαχείριση αποβλήτων και από άλλες χώρες. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσω ποιο είναι το μακροπρόθεσμο σχέδιο. Θέλετε να εξακολουθείτε να ε, αποστέλλετε και να εξάγετε, αν θέλετε, απόβλητα έξω από την Ιταλία ή κάποια στιγμή στοχεύετε να υπάρχει επαρκής ε, ικανότητα διαχείριση αποβλήτων. Και ποιο ποσοστό στοχεύετε να, να αποστέλλετε σε άλλες χώρες εκτός της Ιταλίας. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική συζήτηση αυτή που κάνουμε σήμερα και είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικό που κάνουμε αυτή τη συζήτηση ξανά και ξανά και πάντα μιλάμε για το ίδιο θέμα και βεβαίως είναι σημαντικό. Απλώς θα ήθελα να, με, να έχω στη διάθεσή μου τα ε, έγγραφα εκ των προτέρων, γιατί τώρα μου είναι δύσκολο να καταγράψω όλα αυτά τα σχέδια που μου τα λέτε προφορικά. Θα ήθελα να είμαι σε θέση να προετοιμαστώ για αυτή τη ε, ε, συνεδρίαση και όλοι οι συνάδελφοί μου είμαι ότι το ίδιο θα ήθελαν. Επομένως, αν δεν είναι, είμαστε σε θέση να έχουμε τα έγγραφα εκ των προτέρων, τότε θα πρέπει να αναβάλουμε τη συζήτηση. Και θα πρέπει να είναι εδώ και οι αναφέροντες, όχι μόνο ε, κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Ευχαριστώ. Ε. Ο Τουργκάης, ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Μέρκης. Ε, πρόκειται για μια σημαντική συζήτηση και πολύ σωστά γιατί πριν από λίγες εβδομάδες ψηφίστηκε μια έκθεση σχετικά με τα απόβλητα και ε, ε, για να είμαι και σύντομο όπως ζητάει η Πρόεδρος, θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτη ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε κονδύλια ευρωπαϊκά για να δώσουμε στις περιφέρειες στις για να βελτιώσουν τα πράγματα όσον αφορά τα απόβλητα. Μπορεί να γίνει. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να γίνει, παραλαμβάνω, προς την κατεύθυνση αυτή και κάτι ακόμα. Έχω κάποιες αφιβολίες. Τι γίνεται ποιος στέει ή όχι, η Ιταλική κυβέρνηση ή όχι. Έχουμε φήμες ότι η ιταλικη κυβερνηση οχι εχουμε φημες οτι η επιτροπη ε, θα προσφύγει παραλήψη για τα απόβλητα για την Ιταλική κυβέρνηση. Για πέστε μου, τι γίνεται πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτές τις φήμες. Θα προσφύγει κατά της Ιταλίας επί παραλήψη. Θα γίνει κάτι τέτοιο, ναι ή όχι. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και από μένα μια σύντομη παρατήρηση και μια σύντομη ερώτηση. Άκουσα τις ε, παρατηρήσεις ε, των ε, αναφερόντων και της Κομισιόν. Ακούσαμε για απώλεια της αξιοπιστίας. Η Κομισιόν βλέπει να υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την απελευθέρωση των απαραίτητων πόρων. Τι δυνατότητες βλέπει η Κομισιόν να υπάρχουν ή οι εκπρόσωποι των ε, περιφερειών βραχυπρόθεσμα να ε, μειώσουν ε, το επίπεδο των απορριμμάτων. Η χωρητικότητα είναι περιορισμένη, έρχονται και άλλα απορρίμματα υπάρχουν δυνατότητες βράχη πρόθεσμα με κάποια άμεση στρατηγική να βοηθήσουμε χωρίς χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα. Κανονικά είπε ο κύριος Please, Please. Ωραία, ε, ωραία. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο, διότι βγαίνοντα πριν από λίγο έξω είναι πολίτε, Ευρωπαίοι πολίτε από την Ισπανία που αναμένουν να συζητήσουμε το δεύτερο θέμα και επειδή είμαστε και σε έτος πολιτών μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο και γι' αυτό θα είμαι σύντομο. Δεύτερο, προφανώ ακούσαμε αρκετά πράγματα και θα χρειαζόμαστε να είχαμε μια καλύτερη προετοιμασία μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό έχω παρευρεθεί στη συνεδρία της επιτροπής ε, παρότι δεν ήμουν μέλος να είχαμε και τη γνώμη αυτών που κάνουν αναφορά. δεν ξέρω πώς γίνεται αν έρχονται ειδείς εξόδης δηλαδή με δικά τους έξοδα ή εμείς διευκολύνουμε την παρουσία τους εδώ ώστε να υπάρχει ο αντίλογος. σε αυτά που θα πω με βοηθούν πρώτον αυτά που άκουσα δεύτερο η ιδιότητά μου ως μηχανικού τρίτο η ελληνική εμπειρία καθώς ο παριστάμενος συνάδελφος, ο συνάδελφος Αγκούλο, αναφέρθηκε σε μία έκθεση που πρόσφατα πέρασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων και των απορριμμάτων, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν πάνω από τον μέσο κοινοτικό όρο αναφορών για αυτό το θέμα. Άρα, αρκετά από αυτά που άκουσα από τους εκπροσώπους των αρχών μου θύμισαν ελληνική επιχειρηματολογία, ερώτηση και τοποθέτηση. Γιατί χρειαζόταν τόσες αναφορές για να πάμε επιτέλους σε μια προσπάθεια προσαρμογής στην κοινοτική νομοθεσία, πράγμα που είναι αμφίβολα αν έχει γίνει, καθώς και ο παριστάμενος εκπρόσωπος της Κομισιόν εξέφρασε πάρα πολλές αντιρρήσεις και πάρα πολλές αμφιβολίες. Το δεύτερο, από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Θα μπορούσα και εγώ να μιλάω ώρες εκ της εμπειρίας από αυτών που άκουσα. Το τρίτο, δεν είναι σωστό να δίδονται δημόσια χρήματα, κοινοτικοί προϋπολογισμοί, χρηματοδότησης της τελευταίας και ενδεχομένως έσχατης λύσης αντιμετώπισης των απορριμμάτων όταν το βάρος πρέπει να δοθεί στα πρώτα στάδια κατά τις βέλτιστες πολιτικές που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. Δεν συνεχίζω περισσότερο για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι άλλοι συνάδελφοι. Πιστεύω πως πρέπει οι αναφορές να μείνουν ανοιχτές, να σταματήσει να λειτουργεί από τεφροτήρας, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, να μην δοθούν δημόσια χρήματα, ο φάκελος ανοιχτός μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση σε βάθος όπως ζητούν οι πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Όκεν να ζητήσω συγγνώμη από τους προσκεκλημένους μας, διότι φυσικά κάνουν ό,τι μπορούν. Ε, ε, ακούσαμε και τις παρουσιάσεις τους, αλλά αυτό δεν ε, έγινε με τον τρόπο που συνήθως εργαζόμαστε εδώ πέρα. Συνήθως θα έπρεπε να δούμε τις παρουσιάσεις αυτές γραπτός. Είμαστε η Επιτροπή Αναφορών. Νιώθω άσχημα που δεν έχουμε παρόντες του αναφέροντες. Όταν πρόσφατα το 2010 ε, βρεθήκαμε εκεί. Ε, ακούσαμε ότι λειτουργούν όλα τα συστήματα, αλλά όταν τα είδαμε δεν λειτουργούσαν. Ε, η εγκαταστάσεις για κομποστοποίηση δεν λειτουργούσαν. Θα πρέπει να επισκεφτούμε τα μέρη αυτά αν είναι να δώσουμε το τελικό OK. Πιστεύω θα πρέπει να ακούσουμε τους αναφέροντες και είμαι ικανοποιημένη με την πολύ επιφυλακτική απάντηση της Κομισιόν ε, απέναντι σε αυτά που ακούσαμε. Ελπίζω ε, τα αποτελέσματα να είναι τόσο καλά όσο μας τα παρουσιάσαν εδώ πέρα σήμερα, αλλά θα πρέπει να δούμε πολύ περισσότερα και φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα των φορολογούμενων μας ε, τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε καν αν έχει βγει η μάφια από αυτή την υπόθεση. Πιστεύω ότι πρέπει να κλείσουμε εδώ τώρα, διότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έχουμε ξεπεράσει πολύ το χρόνο μας. Ε, πολύ κακός προγραμματισμός ήταν ο σημερινό ε, και νομίζω θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα τη μέσης διάταξη και να ακούσουμε εκεί του ε, αναφέροντε. Ε, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μάλλον ένα λεπτό για την απάντηση, έτσι. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Συγγνώμη, μόνο για να... μια μικρή παρατήρηση. Επομένω, και ο συνάδελφο αναφέρθηκε σε αυτό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη στη θέση μου ε, για τα κονδύλια. Επομένω, αυτό είναι το ζήτημα το οποίο μα καίει πάντα. Νομίζω ότι η Επιτροπή πολύ καλά κάνει και είναι τόσο αυστηρή και αποδεσμεύει κονδύλια θα αποδεσμεύσει κονδύλια μόνο όταν ε, πληρώσει τις ε, προϋποθέσεις Ιταλία. Ναι, μόνο μια απαντησούλα έτσι από τον εκπρόσωπο της περιφέρειας γιατί είχαμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ναι, ενδεχόμενα γραπτά. Και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, υπέβαλε ένα ερώτημα. Πόσα θα φύγουν από την καμπανία και για πόσο χρονικό διάστημα, τι ποσότητα. Έτσι μπορούμε να τα δούμε μόνο στι διάφορες πτυχές του περιφερειακού προγράμματο. Παρακαλώ τον δόκτωρα Σαντακρότσε. Μια απάντηση άμεση ή μήπως γραπτή λεπτομερική. Αργότερα, μετά, γραπτή. Να σας πω κάτι προκαταρτικά. Ένα λεπτό σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Η Ιταλική κυβέρνηση προβλέπει 150 εκατομμύρια ευρώ. Το ένα μέρος είναι για να ε, μην δυσκολευτεί ιδιαίτερα επειδή δεν υπάρχουν κοινοτικά χρήματα και κάτι ακόμα. Τι περιμένουμε τώρα με εμεί με αυτές τις ε, πρωτοβουλίες και με τη χρηματοδότησή τους τον κύκλο των αποβλήτων να τον φέρουμε σε σταθερό επίπεδο, κανονικό επίπεδο. Θεωρούμε ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα μπορούσαν να κριθούν ε, παραδεκτές, έτσι, δηλαδή να τις δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εμείς η Ιταλική κυβέρνηση σε μας πάει αυτό το κόστος μέχρι να αποδείξουμε ότι αποκαταστήσαμε τον κύκλο το σωστό. Τώρα για τον προορισμό των ε, αποβλήτων. Η Επιτροπή στην έκθεση που δώσαμε μέσω του Προέδρου της περιφέρειάς μας και μέσω της αντιπροσωπείας μας ε, στη Σίταλραπ ε, στις Βρυξέλλες Εκεί χαράξαμε διαγράμματα, βλέπουμε τι γίνεται με την εξαγωγή, την έξοδο αποβλήτων σε εγκαταστάσεις, εργοστάσια άλλων περιφερειών. Οι ποσότητες αυτές έχουν προβλεφθεί όμως στο σχετικό κείμενο έγγραφο. Μπορεί να τα δει κανείς επακριβώς. Βέβαια, επιφυλασσόμεθα να διενεργήσουμε οποιοδήποτε έλεγχο για να μειώσουμε την ποσότητα για την αποστολή εκτός περιφέρειας και τα χρήματα αυτά όπως ε, είπαν ε, και οι δημοτικοί σύμβουλοι που πήραν το λόγο προηγουμένως. Βέβαια με τα χρήματα αυτά χρηματοδοτούμε και τις ε, εγκατάσταση εργοστασίων και ακόμα και χωματερές εκεί που δεν υπάρχουν στο παρόν χωματερές για προσωρινά. Αλλά λοιπόν έχουμε ένα διάγραμμα, στο πούμε έτσι, ροής που δώσαμε στην Επιτροπή. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος Φάλκεμπερκ για απάντηση. Thank you. Um, Σας ευχαριστώ. Δύο συγκεκριμένε ερωτήσεις τέθηκαν. Η μία έχει να κάνει με τη συμμετοχή των περιφερειακών ταμείων. Η γραμμή που έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα είναι ότι μπορούμε μόνο να απελευθερώνουμε οικονομικούς πόρους όταν υπάρχει ένα ε, πρόγραμμα διαχείρισης το οποίο να μπορεί να γίνει αποδεκτό και το οποίο να εφαρμόζεται. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν πολύ προσεκτικά, θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση. Το, το δημοτικό πρόγραμμα μας φαίνεται πολύ καλό και θα δούμε εάν μπορούμε με βάση το πρόγραμμα για τα δημοτικά απορρίμματα να ε, επαναθεωρήσουμε την, ε, την υπόθεση. Βρίσκω όμως δύσκολο να δώσουμε χρήματα από τα Ευρωπαϊκά Διαφθορτικά Ταμεία τη στιγμή που δεν υπάρχουν ε, προγράμματα για την διαχείριση ε, κάποιων απορριμμάτων. Ε, σας είπα στην αρχή ότι μπορεί να μην ε, έχουμε εναλλακτική λύση από το να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Τις επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Ήδη στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς έχει σταλεί η σχετική επιστολή. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας, και τη βοήθειά σας επίσης από τους τοπικούς φορείς, της περιφέρειας και όλα τα όσα πρότειναν. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε και τις γραπτές μνήες αυτό Κλείνουμε τη συζήτηση και όπως ε, ζήτησαν όλοι αφήνουμε ανοιχτές τις ε, αναφορές αυτές. Ναι, αυτά που σας είπα ε, θα σας τα δώσω σε κείμενο ώστε και εσείς να μπορέσετε να τα δώσετε στους υπόλοιπους συναδέλφους σας. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους πολίτες που μόλις ε, εισήλθαν στην αίθουσα. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση με την οποία ξεκινάμε τη συζήτηση αυτών των αναφορών σας. Προχωράμε, προχωράμε αμέσως. Ο πρώτος, ε, ο Ρουπέρες Σαρέγκλη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριοι, κυρίες και κύριοι βοηθοί, καλησπέρα σας. Μισό λεπτό να καταλάβουν τις θέσεις τους όλοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το 3310 για την ασφάλεια στον ενέργειο ισπανικό χώρο και επίσης για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και να πάμε από τα απόβλητα τώρα, να πάμε πετώντας στην Ισπανία και να δούμε το τι κάνουν αρκετοί Ισπανοί, κάτι το ιδιαίτερο επικίνδυνο. Ζητώ συγγνώμη, θα τα πάω τάχιστα, τάχιστα, τάχιστα. Λοιπόν, από τις 16 Ιουνίου του 2011 που και πάλι παρουσιάσαμε τα πράγματα. Είχαμε πάνω από 1.500 καταγγελίες ε, ελεγκτών ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΆΣΑ και Eurocontrol και με αντίγραφο στο ΠΕΤΗ γιατί δεν σέβονται ε, τις μελέτες για την ασφάλεια όπως υποχρεώνει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ρύθμιση πριν από το καινούριο σκηνικό του Ισπανικού νόμου του 2010 του ΕΝΑΤΟΥ. Ακριβώς είχαμε πάνω από 10.000 ε, υπογραφές ε, που δόθηκαν από κυρίως από ελεγκτές ε, σε θέματα ενέργειας ασφάλειας με το νέο πλαίσιο που έθεσε στους ειδικού ελεγκτές το Ισπανικό κράτος και υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις ατυχημάτων και πριν από τις, την ημερομηνία αυτή ακριβώς γιατί όταν υπερίπτανται αεροπλάνα, βλέπουμε ότι πρώτα απ' όλα αντιμετωπίζουν τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και είναι το τρίγωνο ασφάλειας υπηρεσιών ε, αεροπλοείας και ελέγχου. Σύμφωνα με τους κανονισμούς 549-2004, 1108-2009 και 1035-2011. Είναι ο νόμος 2010 και ακριβώς η ερμηνεία που δόθηκε το Μάρτιο του 2001 λέει τι, πώς θα πρέπει να εργάζονται και είδαμε την, υπερ, την υποχρεωτική ημέρα εργασίας που αυξήθηκε η διαρκεία της κατά και 63% σχετικά με το όσο ίσχυαν παλιότερα. Και ακριβώς αυτή η αλλαγή τι σημαίνει σύμφωνα με τον κανονισμό 1035-2011 μια αλλαγή ακριβώς ε, σημαντική στο σύστημα ATM κυρίως των ε, ελεκτή ενέργειας κυκλοφορίας και εκεί στον κανονισμό λέει σχετικά με την ασφάλεια αυτών των υπηρεσιών λέει ακριβώς ότι θα πρέπει πρώτα να γίνουν μελέτες για την ασφάλεια και επιμερισμού των κινδύνων προκαταρτικά πριν να ισχύσει μια αλλαγή από τη στιγμή που θα επηρεάσει το σύστημα ATM. Και ακριβώ στον κανονισμό τη Ευρωπαϊκή πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση πριν από τι αλλαγέ αυτέ, ώστε οι αλλαγέ να μην μειώσουν τη ε, απόδοσή του, ε, το να μπορέσει να αναγνωρίσει τι δύσκολε περιπτώσει κλπ. Δυστυχώς στην Ισπανία δεν ακολουθούμε καθόλου αυτές τις, ε, αυτούς τους κανονισμούς τους ευρωπαϊκούς. Ε, εδώ όλα αυτά έγιναν χωρίς καμία διαβούλευση με τον εργαζόμενο, χωρίς να δούμε τι γίνεται και αναφέρω και πάλι χωρίς να υπάρξουν μελέτες σχετικά με την ασφάλεια και μείωση των κινδύνων για τους ε, ελεγκτές ε, για το νέο πλαίσιο εργασίας τους. Ε, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι τον Ιούνιο του 2011 όταν είχαμε εμφανιστεί και πάλι μπροστά σας ε, η Ούσκα, η Απρόκτα, η Σπίκα, η ΑΠΚΑΕ, η Έτηση Petition ζητήσαμε από τον ΑΕΝΑ ε, και την ΑΕΣΑ να μας διευκολύνουν ε, για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε αυτές τις νέες, ε, αυτούς τους κανονισμούς. Κανείς όμως δεν μας απάντησε ε, ακόμα περιμένουμε πέντε μήνες μετά. Θα πρέπει να σας πούμε εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αυτή η παραβίαση της ρύθμισης της κοινοτική ε, σε παρόμοια θέματα μας βάζει εμάς στην Ισπανία σε μία λεπτή θέση ασυνήθιστη στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ποτέ ένα κρατός ε, δεν κρατήθηκε εγνώση του εκτός από του τριγώνου αυτού ασφαλείας κανονικά όλοι ε, από την πλευρά κυβέρνηση, όσοι ε, υπάρχουν υπηρεσιών, ε, αερογραμμές, πιλότοι, προσωπικό, ελεγκτές, τεχνική συντήρησης, διάφορες εταιρείες, το ένα άλλο, θα πρέπει να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτές τις ρυθμίσεις. Και ακριβώς σύμφωνα με τον κανονισμό 509,4 που είναι ο κανονισμός του ανοιχτού ουρανού όπως είναι γνωστός θα πρέπει σε παρόμοια κατάσταση να παρεύουν γιατί στο άρθρο 13α πρώτα απ' όλα ο στόχος είναι να ισχύουν τα στάνταρτ ασφάλειας στον εννέο ευρωπαϊκό ουρανό και θα πρέπει ε, ταυτόχρονα να αποτρέψουμε κρατημέλη από τα να ακολουθούν παρόμοιες βεβιασμένες διαδικασίες. Ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ε, μέλη της Επιτροπής Αναφορών, να σας πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε το έργο μας έτσι, γιατί ε, υπάρχει πιθανότητε για ένα αεροπορικό ατύχημα. Σύμφωνα με τον κοσμό 1035-11 στο παράρτημα 1, ο πάροχος υπηρεσιών παρομοίων θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπογράψει ότι είναι υπεύθυνο σύμφωνα με την κατάσταση που ισχύει από νομικής πλευράς. Δηλαδή, κάλυψη ότι ναι, ψεύεται κανείς το νομικό πλαίσιο του ενιαίου ανοιχτού ουρανού. Δεν συμβαίνει όμως αυτό στην Ισπανία και για άλλους λόγους ε, δεν υπάρχει πραγματική ανάπτυξη, ε, υπάρχει φόβος, πανικός, γιατί πολλές φορές απειλούνται με απόλυση οι ελεγκτές ε, και αναλαμβάνουν έργο πολύ πιο βαρύ και πολύ περισσότερο από συνηθίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παντού όλοι διαμαρτύρονται, όλοι θέλουν να γίνει σεβαστή αυτός, αυτός ο ανοιχτός, ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός δεν θα πρέπει να αποσιωπήσουμε ότι έχει ροτερεύσει η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια την εναέρεια στην Ισπανία. Ε, γιατί αυτό είναι εδώ μια δικτατορία, δικτατορικά μέτρα, χωρίς νόημα, γιατί δεν απαντώνται ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και είναι δύσκολη η κατάσταση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες της ασφάλειας. Έτσι, just culture, έτσι τα γνωρίζουμε. Γιατί με διάφορες μελέτες τα αυτά τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι επειδή το Ισπανικό κράτος δεν συζητάει με τους ε, ελεκτές ενεργή κυκλοφορίας, βλέπουμε ότι ακριβώς μαθηματικά έχει αυξηθεί ο κίνδυνος κατά ένα ανισχυτικό 75%. 75% περισσότερος κίνδυνος. Ε, καταλαβαίνετε ε, τι γίνεται. Κανείς δεν παρεμβαίνει, κανείς δεν βελτιώνει. Ακριβώς και διαφορετικά θα πρέπει ακριβώς ο Ευρωπαϊκός Νόμος να κηρύξει την Ισπανία, τον ενέριο, το φύρ της Ισπανίας σαν ένα υποχώρο του ανοιχτού του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού χωρίς την απαιτούμενη ασφάλεια. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείε διατρέχουν κινδύνους ε, σε περίπτωση κινδύνου, ατυχήματος και λοιπά, λόγω της πλημερούς, ε, του πλημελούς ελέγχου δεν μπορεί να αποδοθεί στους ελεγκτές. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πρωτοφανής κίνδυνος από τότε που μέσω της Συμφωνίας της Βαρσοβίας ε, υπεγράφηκε η συμφωνία αυτή. Άρα λοιπόν ε, ε, μην ξεχνάμε ότι παλιότερα είχαμε ένα τρομερό εμπορικό ατύχημα σε εμπορικό αεροπλάνο μεταφορών. Ε, μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρξει ο διάλογος. Θα πρέπει να σεβαστούν και τον εθνικό νόμο και τον κοινοτικό νόμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Φορέας θα πρέπει να εργαστούν και μαζί με τους επαγγελματίες στην Ισπανία, οι οποίοι επαγγελματίες, οι ελεκτές αυτοί θα μπορέσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια στον εναέριο ισπανικό χώρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρουιθ Πέρεθ και ο αναφέροντα τον αναφέροντα Χίλ Παρακαλώ, μην ε, μακρηγορήσει. Όχι, όχι, λάθος. Ε, δεν είμαι ο προηγούμενος, είμαι επόμενος. Ναι, κύριε Τονγκάης. Κυρίες και κύριοι, η Συνδικαλιστική Ένωση η εγώ είμαι πρόεδρος της. Ε, το 2010 ήρθαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό για να καταγγείλουμε τα όσα γίνονται σε ένα Ευρωπαϊκό που ανησυχούσε Παρακαλώ, παρακαλώ, μην, τρέχετε τόσο, δεν σας, δεν σας προλαβαίνουμε. Οι διερμηνείς μας ε, δυσκολεύονται άσχημα. Ναι, εντάξει, εντάξει, αλλά και εσείς δώστε μου λίγο χρόνο. Ναι, ναι, θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, και εντάξει, δέχτηκαν και μείωση μισθού, ε, κατά 50%. Άρα λοιπόν ε, να είμαστε φερέγγοι είπαν ε, και τώρα είμαστε με την αρμόδια υπουργού που είπε ότι από 200 εκατομμύρια ε, μάλλον έχουν αυξηθεί εντελώς τα νούμερα, η μισθή, το ένα το άλλο και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το πώς επηρεάζει ο μισθός μας, πόσο λίγο επηρεάζει ο μισθός μας το σχετικό, ε, τη σχετική ζημιά. Εδώ θα πρέπει ηθικά, επαγγελματικά να μην ξεχνάμε το τι γίνεται. Υπάρχουν πολλοί που δεν προλάβαιναν ε, και εδώ, στον ίδιο χώρο αυτό, καταγγείλαμε τις δυσκολίες μας. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση για τους ελεκτές εναερές κυκλοφορίας Ισπανίας. Είχαμε 200 εκατομμύρια ε, ταξιδιώτες ε, το, πέρυσι ε, που πέρασαν από τον χώρο μας, αλλά είχαμε 47 σχεδόν συγκρούσεις και 95 ατυχήματα, μικροατυχήματα το 2010. Ενώ στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, δεν είχαν 47 και 95, είχαν 0 και 0. Ε, καταλαβαίνετε το Eurocontrol τι λέει, ότι έχουμε στην Ισπανία το 5% της κίνησης της ευρωπαϊκής και 50% των παραβιάσεων, ε, παραβάσεων. Ε, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι αντιστοιχούν στην αλήθεια, αντιστοιχούν σε όσα είχαμε πει και στο παρελθόν. Ε, έχουμε εδώ τις δύο ας πούμε παραβάσεις σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 1035-2011 ακριβώς οι πάροχοι υπηρεσιών θα προσπαθήσουν όμως, λέει ο κανονισμός, να βελτιώσουν την κατάσταση μέσω των κατάλληλων μηχανισμών. Ε, βλέπετε τι έκανε όμως η ένα σχετικά με τον κανονισμό αυτό. Και το δεύτερο που εμφανίζεται σε αυτόν τον κανονισμό λέει ότι Safe Management Systems ε, αυτό ε, θα έχει ακριβώς ε, την απόλυτη προτεραιότητα που θα αποδώσει σε την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επίπεδου μεταφοράς και δυστυχώς η κατάσταση καθόλου μα καθόλου δεν άλλαξε. Καταλαβαίνετε ότι και το προσωπικό υποφέρει από τη διοίκηση που δεν ακούει κανέναν, ούτε επαγγελματία, ούτε έχει καμία διάθεση να διαπραγματευτεί. Δεν το λέω εγώ αυτό, το είπε ο προηγούμενος πρόεδρος της ΑΕΝΑ που είπε στο ΕΛΠΑΙΣ ότι το μεγαλύτερο ακριβώς λάθος του ήταν ότι οι αλλαγές στην ΑΕΝΑ δεν έγιναν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς η ΑΕΣΑ κανονικά που θεωρητικά εγγυάται την ασφάλεια την ενέργεια, ε, τι έκανε ε, και έκρυψε αυτά τα στοιχεία αλλά ταυτόχρονα προσπάθησε να ενοχοποιήσει τους ε, ελεκτές. ίδια ε, αποφάσιζε και είπε ότι το 20% των ελεκτών είναι ένοχοι και κινδυνεύουν με πρόστιμα από 90.000 έως 225.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, δεν σας προλαβαίνουν, δεν σας προλαβαίνουν. Ναι. Ε, η ίδια αποφασίζει, η ίδια καθορίζει και τα πρόστιμα, καταλαβαίνετε. Εδώ ε, Κανονικά θα έπρεπε όμως να κάνει και μια κάποια έρευνα για τους πάροχους υπηρεσιών και όχι για το προσωπικό. Ε, βλέπουμε ότι παραβιάζει το 4,2 του 1035 του 2011 άρθρο που λέει ότι η αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει ακριβώς αν όλα αυτά γίνονται σεβαστά πριν να δώσει σε κάποιον ένα πιστοποιητικό ώστε να γίνει υπάρχος υπηρεσιών. Βλέπετε ότι ταυτόχρονα η προηγούμενη κυβέρνηση τι πονηρά έκανε. Γιατί ε, όλες αυτές ε, οι κατηγορίες για παραβάσεις κλπ. πότε τις υπέγραψαν 19 Νοεμβρίου πέρυσι ακριβώς την παραμονή των εκλεγών ήξερε η κυβέρνηση ότι θα χάσει τις εκλογές και το έκανε δωράκι δηλητηριασμένο δωράκι στην επόμενη κυβέρνηση τότε που ε, δόθηκαν υπογραφές αυτό έγινε το Σάββατο κανονικά είναι κλειστά το Σάββατο Άρα λοιπόν τους κοινοποιήθηκαν αυτές οι παραβάσεις ε, τη Δευτέρα, όταν ακριβώς ε, είχαν βγει τα αποτελέσματα των εκλογών της 20 Νοεμβρίου. Βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά που έχουν γίνει. Όλα αυτά τα προμελέτησαν και θέλησαν να υπονομεύσουν την καινούρια κυβέρνηση που προήλθε από τις εκλογές. Αλλά εδώ ακριβώς ε, τι βλέπουμε, ότι αυτοί οι ίδιοι οι ελεγκτές υποφέρουν ε, και κινδυνεύουν ε, να κλειστούν και στις φυλακές γιατί μια κάποια μέρα ε, έκλεισαν τον εναέριο χώρο της Ισπανίας γιατί είπαν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται, ε, πώς, πώς, πώς, πώς κάποιοι που δεν θέλουν να δουλέψουν ακριβώς επειδή υπάρχει κίνδυνος, πώς κατηγορούνται ότι δεν σέβονται τις προδιαγραφές. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, η προηγούμενη κυβέρνηση δημιούργησε αυτό το κλίμα, ώστε η σημερινή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα αξεπέραστο σχεδόν πρόβλημα. Αυτό και γίνεται. Σας το έλεγα λοιπόν ότι δεν σέβονται τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους κανονισμούς. Όλα αυτά μας προκαλούν ντροπή. Έτσι, λοιπόν, ε, όλα αυτά που δεν σέβονται είναι πολλά και διάφορα. είναι σαν ένα κρεμμύδι που σιγά σιγά του βγάζουν τα στρώματά του. Στο τέλος δεν μας μείνει τίποτα από το αρχικό κρεμμύδι. Εδώ η σχετική μελέτη δείχνει ακριβώς ποιοι φταίνε και σας, ε, θα σας δώσω την έκθεση αυτή. Και κανονικά πρέπει να μιλάμε για επίπεδα ασφάλειας. Σας είπα προηγουμένως ε, για το κρεμμύδι αυτό, του αφαιρούνται σιγά σιγά στρώματα και δεν θα μείνει τίποτα, ένας τρομερός μεγάλος κίνδυνος. Εμείς εργαζόμαστε όσο γίνεται με πιο επαγγελματικό τρόπο για να πετύχουμε. Και ευτυχώ να είναι καλά, δηλαδή δόξα τω Θεώ λέει ο μιλήτης, τα καταφέρνουμε προς το παρόν, αλλά μέχρι πού θα πάει αυτό. Εμείς ελπίζουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σωστά, γιατί διαφορετικά η μόνη ικανοποίηση που θα μας μείνει μετά από ένα τύχημα ότι εμείς το είχαμε προβλέψει, το είχαμε αναγγείλει ουσιαστικά. Έτσι, σε όλου του χώρου, ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είστε όλοι εκπλεγμένοι από τη λαϊκή βούληση. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε την κατάσταση. Όπως σας είπα, σας δίνω την έκθεση με διάφορα θέματα, σύμφωνα και με το σχετικό ισπανικό νόμο. Όλα αυτά είναι κατά της εναέριας ασφάλισης, ασφάλειας και κατά των πολιτών. Εδώ όλα αυτά τα στοιχεία ε, είναι απαράδεκτα, είναι απαράδεκτα. Τι γίνεται αλλού σε άλλα κράτη-μέλη, σύμφωνα και με τις στατιστικές του Eurocontrol, σέβονται ως αυτές τις ρυθμίσεις. Εμείς όχι. Ε, όχι εμείς ε, όσοι τα ρυθμίζουν αυτά. Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια. Αυτή είναι και το κλειδί μιας σωστής δουλειάς για αυτά. Ε, θα πρέπει να πετούν ε, ασφαλείς οι πελάτες μας. Μπεατρίστο Τόμας. Ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να απαντήσει σε όλα όσα επόθηκαν και πάλι ε, το ζήτημα αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί. Ε, σήμερα οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας ε, αναφέρθηκαν σε ζητήματα που έχουν επαναλάβει πολλές φορές. Ε, και αναφέρθηκαν σε κατηγορίες που δυστυχώς δεν μπορούν να στηριχθούν από αδιάσυστα στοιχεία, δηλαδή μη συμμόρφωση με της ε, Ισπανικής νομοθεσίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές ε, στον ενιαίο εναέριο χώρο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση της Ισπανικής νομοθεσίας. Όπως ε, ε, ανέφεραν και οι αναφέροντες, και όπως ανέφερε και το δικαστήριο, το ζήτημα αυτό είναι αρμοδιότητα της εθνικής νομοθεσίας. Υπόκειται στην εθνική νομοθεσία λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενέργεια ασφάλεια. Ακόμα και αν είναι κάτι για το οποίο δεν είμαι αρμόδια, εφόσον εγώ ε, εργάζομαι στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας κυκλοφορίας, οι αναφέροντες μας ζήτησαν να ζητήσουμε από την ΑΕΝΑ για να ε, εκπονήσει μία έρευνα επιτόπου. Εμείς μαζί με τους αδέλφους μας της ενέργειας κυκλοφορίας ε, παρατηρήσαμε το έργο της ΕΑΖΑ Και δεν είναι η Ισπανία με τις χώρες ε, που αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΑΣΑ, γιατί εκεί από τις προτεραιότητες αποτελούν οι χώρες όπου η ασφάλεια στις χώρες όπου υπάρχουν περισσότερες απειλές ε, για την ε, ενέργεια ασφάλεια. Ωστόσο, η ΕΑΣΑ είπε ότι μπορεί να επιδείξει ευελιξία ε, και κατόπιν αιτήματο της Επιτροπής θα μπορούσε να εκπαιδεύσει διοικητική έρευνα. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θα ήθελε η ΕΑΣΑ να αποτελεί αντικείμενο χειραγώγησης από τις Ισπανικές αρχές. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, πολλές από αυτές τις κατηγορίες αφορούν ε, το εθνικό δίκαιο και ε, το να αναφερόμαστε στο κοινοτικό δίκαιο εκεί που δεν πρέπει θα μας οδηγήσει σε προβλήματα. Εξάλλου, η ΕΑΣΑ έχει αρκετά ευέλικτο πρόγραμμα για να μπορέσει να επιτρέψει μια τέτοια διοικητική έρευνα. Ευχαριστώ. Η πρόεδρο σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μπουστινάρου. Μπουστινάρου. Ευχαριστώ. Να μιλήσω ρουμανικά. Θα μιλήσω στα ρουμανικά γιατί εδώ έχουμε ιδιαίτερα τεχνικά ζητήματα και ζητήματα θεμελιώδη για την ασφάλεια της ενέργειας κυκλοφορίας και των ενέργειων μεταφορών στην Ισπανία. Αρνούμε να δεχθώ ότι ένας, μια οργάνωση που εκπροσωπεί τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας στην Ισπανία πέτυχε να κινητοποιήσει χιλιάδες ανθρώπων κάτι που προηγουμένω δεν είχε επιτευχθεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό ε, έγινε μόνο για λόγους ε, των σωματείων, συνδικαλιστικού αν θέλετε. Όμως δεν συμφωνώ με την Επιτροπή. Δεύτερον, στην αναφορά τους ε, η Ένωση αναφέρεται σε στατιστικά στοιχεία που υπογραμμίζουν τους κινδύνους ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στις ενιαίε μεταφορές στην Ισπανία. Κανένας από εμά δεν είναι εμπειρογνώμων ειδικό στην ενιαία ασφάλεια. Επομένως, θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ισπανική κυβέρνηση να μας ενημερώσει μέσω επισήμου εγγράφου το στομότερο δυνατόν και όταν λέω το στομότερο δυνατόν, ε, εννοώ με όρου του Κοινοβουλίου, δηλαδή να μας ενημερώσει η κυβέρνηση εάν τα όσα αναφέρουν οι αναφέροντες ισχύουν ή όχι. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από την Επιτροπή Είπατε ότι η εναέρια ασφάλεια είναι πρόβλημα της ισπανικής κυβέρνησης, όμως η ενεργεια ασφαλεια ειναι προβλημα της νομοθεσίας και ο τρόπος λειτουργίας, το modus operandi, θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα και τη επιτροπή, όταν ε, υπάρχουν προειδοποιήσεις για συγκεκριμένους κινδύνους που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να θίξω. Εδώ δεν μιλάμε για κοινωνικά δικαιώματα. Παρόλο που υπάρχει αναφορά σε κοινωνικά δικαιώματα εδώ, Νομίζω ότι το θεμελιώδες ε, στοιχείο ε, της αναφοράς είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια στις ενέργειες μεταφορές και πτήσεις για τα 200 εκατομμύρια επιβατών κάθε χρόνο. Εάν η Επιτροπή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης ΜΟΥΒ και η Ισπανική Κυβέρνηση μπορούν επισήμως να μας καθησυχάσουν ότι πληρούνται όλα τα πρότυπα και ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι, τότε μπορούμε και εμείς ε, να θέσουμε αναμφιβόλο το, τα αιτήματα των ε, αναφερόντων. Ε, τέλος, θα ήθελα το αίτημα των αναφερόντων να μείνει ανοιχτό έως ε, ότου μας ε, παρασχεθούν τέτοιες σαφείς και ξεκαθαρές απαντήσεις. Εξετάζω επίση το ενδεχόμενο να στείλω αυτή την αναφορά στην Επιτροπή Τραν, Επιτροπή Μεταφορών, για να μπορέσουν και οι συνάδελφοι να ε, επαληθεύσουν ε, την ισχύ των στοιχείων ε, της αναφοράς και το κατά πόσο η αξιολόγηση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στις προσδοκίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, άκουσα τους, συναδέλφους, τους ε, ε, αναφερόμενους. Θέλω να μιλήσω εκ μέρους της ΓΚΟΕ, αλλά κυρίως θέλω να μιλήσω εκ μέρους του συναδέλφου του κυρίου Μέγερ, ο οποίος για εκτάκτους λόγους δεν είναι παρόν εδώ. Έχουμε κάνει συνεργασία όμως, με έχει ενημερώσει, άκουσα και τους αναφερόμενους. Πρώτο, αναδεικνύεται μείζον θέμα ασφάλειας των πτήσεων. Και ρωτώ την εκπρόσωπο της Επιτροπής, αν τα στοιχεία που μας δίδουν οι ενώσεις των ελεκτών είναι αμφισβητούμενα. Ρωτάμε, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας, ισπανικές αρχές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μας δώσει τα ακριβή και συγκεκριμένα στοιχεία. Διότι, αν είναι σωστό, το έχω αυτό το στοιχείο, το ανέφεραν και οι εκπρόσωποι των ε, ελεκτών, στην Ισπανία με το 5% της κίνησης όσο αφορά τις εναέριες επικοινωνίες στην Ευρώπη έχουμε πολλαπλά γεγονότα τύπου ατυχήματος από τις άλλες χώρες τότε ή δεν είναι καλά, δεν μας δίνουν αληθινά στοιχεία, ή εκεί δεν μπορούν να οδηγήσουν καλά τα αεροπλάνα, ή κάτι άλλο γίνεται. Και επειδή ξέρουμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, η λογική συνέπεια είναι ότι κάτι γίνεται που σημαίνει ότι η νομοθεσία που έχει επιβληθεί έχει εντατικοποίησει τη δουλειά και έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση στον εναέριο χώρο της Ισπανίας έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Το δεύτερο, πάλι απευθύνομαι στην εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ποια σημεία ακριβώς από αυτά που αναφέρονται δεν εμπίπτουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ενδεχομένως, επειδή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία μπαίνουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη των δικαιωμάτων ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά. Το δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη να μετακινείται με ασφάλεια τουλάχιστον στους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Έχει στοιχεία όλων των προηγουμένων, ενδεχομένως είναι δικαίωμα νέου τύπου, άρα η ευρωπαϊκή νομοθεσία ή πρέπει να προσαρμοστεί ή πρέπει να βρει τις γενικές αναφορές για να συναντήσουμε αυτό το δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί κάπου με λεπτομέρειες δεν περιγράφεται ότι υπάρχει το δικαίωμα εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες να περνάμε με ασφάλεια από τον εναέριο χώρο της Ισπανίας. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γιατί ήδη έχει εξαντληθεί ο χρόνος. Νομίζω ότι πρέπει να μας δοθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία, να μείνει ανοιχτό να ψαχτεί καλύτερα το θέμα. Δεν θα ήμουν αντίθετο με την πρόταση του κυρίου συναδέλφου να απευθύνουμε τη σχετική αναφορά και στην Επιτροπή Μεταφορών, αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να διαφορούμε είτε θεωρώντας ότι είναι ένα ισπανικό πρόβλημα, είτε θεωρώντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και τα στοιχεία και ούτε καθεξής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Μαρτίνες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι. ναι, θα μιλήσω για ένα προσωπικό μου λογαριασμό. Ε, εμένα θα εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άκουσα αυτά που είπε η Επιτροπή μου και ο Γενικός Διευθυντής του Eurocontrol που μας είχε καλέσει και ε, τι γίνεται εδώ πέρα, γελιοποιούμεθα εδώ στην Επιτροπή ε, Αναφορών. Εμείς θα έπρεπε να ξέρουμε πριν να καλέσουμε το Eurocontrol τι ακριβώς απαντάει ακριβώς, ε, τι συμφωνεί, τι όχι. Και όλα αυτά, αν αφορούν το Eurocontrol, να έχει κάτι να μας πει, τι γίνεται εδώ. Από ό,τι λέει εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω από το Γενικό Διευθυντή, δεν έχω τίποτα να πω αλλά με την προηγούμενη κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώ είναι κράτο δικαίου η Ισπανία, έτσι. Έτσι τουλάχιστον το χαρακτηρίζουμε. Δεν νομίζω να το αφισβητεί κανεί τώρα. Αυτό ισχύει. Και αυτό ότι δίθεν παραβιάσει πάνω στην ισπανική νομοθεσία. Αυτά τα πράγματα δεν τα συζητάμε ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε στην Επιτροπή Αναφόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν έχει άλλωστε και την αρμοδιότητα να ασχοληθεί με παραβίαση νομοθεσίας κράτους μέλους. Εντάξει, να διατηρηθεί ανοιχτή αναφορά, γιατί όχι. Γιατί κάτι που μας ανησυχεί σίγουρα θα πρέπει να σημάνει συναγερμό. εντάξει, θα πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτή όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, να δοθούν εξηγήσει εκεί που απαιτούνται αυτές οι εξηγήσει και να καταλάβουμε το τι γίνεται. Και άλλωστε εμεί οι ίδιοι πετάμε και πετάμε και ξαναπετάμε περισσότερο <laughs> και αρκετοί από εμά και του Ισπανου. μάλιστα παραπετάμε εκεί πάνω. Λοιπόν, εάν ε, ισχύουν αυτά ότι υπάρχει τρομερός κίνδυνος θα πρέπει να αλλάξουμε και μέσο μεταφοράς. Να πηγαίνουμε πια με αεροπλάνο, να πηγαίνουμε με άλλο μέσο. Αυτό λοιπόν ισχύουν όλα αυτά που υποστηρίζουν. Εντάξει, αν το σκέφτονται έτσι, αν ε, διατηρούν τη θέση τους, αλλά να πάνε εκεί που είναι οι αρμόδιοι για να αποφασίσουν και όχι αλλού σε άλλους χώρους που δεν υπάρχουν αρμόδιότητες. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα που υποστηρίζονται μήπως είναι απλά εσκεμένα για να αλλάξουμε μία νόμιμη ανησυχία, να την πάμε σε άλλο τομέα, λέγω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ο Τουργκάης. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Από Μαρτίνεθ αυτό του Προέδρου του Eurocontrol. Τι γίνεται εδώ. Γιατί δεν μας απαντήθηκε όπως πρέπει. Εδώ με έχει απογοητεύσει όταν είχαν έρθει εδώ οι αναφέροντες και τώρα, ξαν... Ε, και τώρα επέστρεψαν. Είχαμε ζητήσει να μας ενημερώσει το Eurocontrol και να μας δώσουν πληροφορίες πάνω στην υπόθεση αυτή. Τώρα γιατί δεν ενδιαφέρθηκε, δεν ήθελε έτσι, δεν έχει αρμοδιότητα, τι ισχύει εδώ, γιατί. Αλλά από τη στιγμή που ζητάμε ασφάλεια, εναέρια ασφάλεια, θα πρέπει να μπορούμε να ακούσουμε τους αρμόδιους και γι' αυτό ακριβώς. Αυτό δεν το πετυχαίνουμε σήμερα. Δεν ακούμε αυτό που θα έπρεπε να μπορέσει να πει το Eurocontrol και εδώ μπροστά στους αναφέροντες και στην δικιά μας την Επιτροπή Αναφορών την ίδια. Με τα θέματα αυτά επειδή ο κύριο Μποστινάρου έθεσε ένα θέμα, παραμένει είπε να παραμείνει ανοιχτό και εκείνο και να ζητήσουμε περισσότερε πληροφορίε για να δούμε, να προσθεθούν σε όλα αυτά που διαθέτουμε. Εντάξει, κανένα πρόβλημα να παραμείνει ανοιχτό και ναι, ζητάω να διατηρηθεί ανοιχτό, ανοιχτή αυτή η αναφορά. Α τουλάχιστον στο Eurocontrol να στείλουμε ένα σημειωματάκι και να πούμε ότι μας απογοήτευσε το ότι δεν απαντάει το Eurocontrol στην Επιτροπή μας Αναφορών. Σας ευχαριστώ. ΟΚΕΝ Θα είμαι πολύ σύντομη. Να σας ενημερώσω ότι θα ρωτήσουμε την κυβέρνηση και να σας πω επίσης ότι η ότι έχουμε και την πρόταση της Επιτροπής να συμμετάσχει και η υπηρεσία και νομίζω θα πρέπει να δεχτούμε ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας να ασχοληθούμε με το θέμα. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες και οι πολίτες μας ενδιαφέρουν, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να απαντήσουμε με τρόπο αξιοπρεπή. Θα ε, έπρεπε να έχουμε θεωρήσει ε, απαράδεκτη την, ε, την αναφορά εάν ε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε του προσκεκλημένου ε, και να κλείσουμε εδώ το θέμα, διότι ε, ήδη έχει περάσει μισή ώρα παραπάνω από ό,τι είχαμε. Μια απαντησούλα, μια απαντησούλα. Ένα λεπτό, εντάξει. Ένα λεπτό απάντηση. Ποιο εσύ, εγώ. Μισό λεπτό. Ακριβώς εκεί που έπρεπε. Αυτό είπε ο κ. Μποστινάρου. Είχαμε πει και ξεκινώντα από αυτά συναντήσεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μας πετάνε το μπαλάκι από τι κοινωνικές υποθέσεις, από τα θεμελιώδη δικαιώματα, από τις μεταφορές, ε, μας πηγαίνουν φέρνουν. Κάποιος από, από το γίγο της κυρίας ε, Ρέντιν ε, κάθε τόσο μας λένε είναι από εδώ, από εκεί, από παρακάτω, μεταφορές, αναφορές και μας πάνε και στις κοινωνικέ υποθέσεις. Και τώρα σήμερα στη μέση για διάταξη εδώ, σαν να είμαστε για τις κοινωνικέ υποθέσεις. Είναι θέμα εναέριας ασφάλειας. Κύριε Μαρτίνες, δεν θα απαντήσω, είναι απόν, αλλά τέλος πάντων, να απαντήσω. Δεν έχει ιδέα τι του γίνεται. Εδώ πέρα δεν ξέρει τι γίνεται με την εναέρια ασφάλεια. Ο ενίος ευρωπαϊκός ουρανός πάει παραπέρα από τα εθνικά σύνορα. Υπάρχουν πάρα πολλέ ρυθμίσει, κανονισμοί και θα πρέπει να του σεβαστούν αυτού του κανονισμού από την πρώτη μέρα δημοσίευσή του, κοινοποίησή του. Εντάξει, και ότι λένε ότι είναι κυριαρχό κράτο η Ισπανία, άρα λοιπόν δεν πρέπει να κατεβόμαστε και κράτο δικαίου. Κράτο δικαίου και μα μας βάζει σε στρατιωτικό καθεστώ και μα βάζει το πιστόλι στον κρόταφο και μα λέει αυτά είναι, έτσι θα εργαστείτε. Αυτό είναι το κράτο δικαίου που υποστηρίζει ο κύριο Μαρτίνεθ ότι ισχύει στην Ισπανία. Όχι, δεν είναι αυτό. Εντάξει, και ο συνάδελφος εδώ πέρα, θα, αν μπορεί να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, με επιτρέπετε, με επιτρέπετε 20 λεπτά. Μια ερώτηση. Σημαντικό είναι. Πριν να μιλήσει ο τελευταίος. Μπορείτε να μας πείτε για να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι βουλευτέ. Γιατί στις κοινωνικές υποθέσεις και όχι στις μεταφορές ή ασφάλειας. Είναι σημαντικό να μας το πείτε κι εσείς. Πού, πού, πού, ποια, ποιανού δικαιοδοσία τελικά δηλαδή. Πού το πάτε εσείς. Ε, πράγματι όταν παρουσίασαν την αναφορά τους οι αναφέροντες βασίζονταν στο, στην ισπανική νομοθεσία που μείωνε για εκείνους ε, την δυνατότητά τους να εργάζονται με υπερορίες. Ε, αυτό μπορεί να επηρεάσει το δικαίωμα στην εργασία τους και γι' αυτό θεώρησαν ότι οι ώρες ήταν ουσιαστικά καταναστική εργασία. Ε, και αυτό αντιβαίνει στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε ορισμένα άρθρα ε, της συνθήκης. Γι' αυτό και αυτή η αναφορά αρχικά απευθυνόταν στην Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, μετά η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών MOVE ε, συνέβαλε στη συζήτηση και όταν η κυρία Ρέντινγκ εξήγησε ότι αυτά τα στοιχεία δεν μπορούσαν να οδηγήσουν στο χαρακτηρισμό της εργασίας ε, των ελεγκτών ως καταναγκαστικής εργασίας, αλλά θα μπορούσαν να επηρεάσει τις ενέργειες μεταφορές. Αυτό το στοιχείο το αξιοποίησαν οι αναφέροντες για να, ε, ε, να αλλάξουν κατεύθυνση προς αυτό το ζήτημα της εναρίας ασφάλειας. Και η ήταν η ίδια αναφορά με τον ίδιο αριθμό. Επομένως, ε, από κοινωνικής πλευράς απαντήσαμε αρνητικά γιατί αφορά, είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας και έτσι μετακινήθηκε. Αν όμως θεωρούμε ότι πάει προς άλλον τομέα αλλά κρατάει τον ίδιο αριθμό, δηλαδή για άλλο θέμα αλλά για τον ίδιο αριθμό, τότε θα τύχει εξέταση ε, και από τις Γενικές Διεύθυνσεις ε, Απασχόλησης και Γενικές Διεύθυνσεις Μεταφορών. Ε, επομένως, ε, εξετάσαμε και το Βασιλικό Διάταγμα 5-2010 και 9-2010 και δεν έχουμε βρει μέχρι τώρα καμία συμβατότητα με την Εθνική Νομοθεσία. Και μπορώ να καθησυχάσω ε, τα μέλη της Επιτροπής αυτής ότι εάν υπάρχει ένα στοιχείο που επηρεάζει την ενιαία ασφάλεια στην Ισπανία σε σύνδεση βέβαια και ε, με τους σενάριους χώρους άλλων κρατών μελών. Βεβαίως και η Επιτροπή θα ε, εξέταζε το ζήτημα για να το ρυθμίσει είτε στο εσωτερικό της ε, Επιτροπής Ενέρας Ασφάλειας είτε βάσει του μαύρου καταλόγου της ίδιας Επιτροπής. Και η Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνε έναν αέριο χώρο έξω από τις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ε, Για να τελειώσουμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο κ. Μποστινάρου πρώτα. Μία και μόνο παρατήρηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσουμε όλες αυτές τις στοιχές. Γιατί όταν κάποιος ε, ενώπιον του Κοινοβουλίου αναφέρει προβλήματα που συνδέονται με την ενέργεια ασφάλεια. Ένα από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με το, ένα από του μεγαλύτερου αριθμού επιβατών επί έτος, θα πρέπει κατευθείαν να το ε, επιλύσουμε για, να, για, και για την αξιοπιστία τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ζητημάτων που άπτονται τη ασφάλεια. Για να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Μποστινάρου, διακόπτεται ο μιλητής. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ε, πολιτών, ε, συμμερίζουμε πολύ το στην άποψή σας. Αν με οποιοδήποτε τρόπο ε, διακινδυνεύεται η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών, προφανώς και ο ισπανικός εναέριος χώρος θα αποκλειόταν, θα έκλεινε. το έχουμε έναν, είχαμε έναν αξιωματούχο όπως network operator θα είχαμε, αν υπήρχε πραγματικό πρόβλημα, θα είχαμε και καταγγελίες από πολίτες, αλλά αυτό δεν ισχύει. Σε 10 δευτερόλεπτα να... δέκα δευτερόλεπτα να απαντήσω ο κ. Κοπεστινάρου και εδώ δίπλα λυπάμαι, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω το όνομα. Performance Review Report έτσι από πλευρά Eurocontrol είναι του 2010, είναι επίσημες εκθέσεις, είναι στο σελίδα του Eurocontrol και σελίδες από τους πάροχους υπηρεσιών εκεί και από εθνικούς ε, και κανονικά τον Ιούνιο έπρεπε να το έχω, το έφερα τώρα αλλά τα 2010 έχουμε 47 τύπου α σχεδόν ατυχήματα και 50 τόσα β. Ενώ φέτος ε, είναι, ταυτίζονται με τις ευρωπαϊκές στατιστικές οι ισπανικές αυτή τη χρονιά. Τι γίνεται, γιατί αυτή η διαφορά. καμία άλλη παρέμβαση, το είπε και ο Στάφος Μαρτίνες. Πάνω στο θέμα αυτό δεν μπορούμε να τα πάρουμε έτσι ελαφρά την καρδία πέρα από τις ειδικέ αρμοδιότητες. Κυρία ζητάει το λόγο και πάλι. Ναι, αν θέλετε, λοιπόν, εσάς ευχαριστώ. Για το PRB, για την έκθεση αυτή, είχαν την draft ε, όταν το PRB ακριβώς ε, υποβάλλει ένα σχέδιο έκθεσης για θέματα εναέριας ασφάλειας. Η πρώτη έκθεση που πάει σε εθνικές αρχές, σε όλα τα κράτη-μέλη, ο καθένας για εκείνο που τον αφορά. Θα πρέπει να διορθώνονται τα στοιχεία, να ξεκαθαρίζουν ε, από ορισμένα στοιχεία που δεν τα έχει υπερμπέ. Και από τη στιγμή που απαντήσουν τα κράτη-μέλη, τότε διορθώνεται αυτή η έκθεση και μάλιστα με τον τρόπο τον πρέποντα. Όταν έχουμε μετά την τελική έκθεση για την Ισπανία που δημοσιεύτηκε, αυτά τα 47 τύπο α σχεδόν ατυχήματα που λένε οι αναφέροντες, δεν υπήρχαν αυτά τα 47. Αυτά και ευχαριστώ. Ε, ε, ε, εντάξει, εντάξει και εμείς θα εκτιμήσουμε στο κάτω-κάτω, στο τέλος-τέλος ας πούμε να δούμε όλα αυτά που ακούσαμε και μετά να πάρουμε και την απόφασή μας. Λοιπόν, όλοι οι συνάδελφοι είπαν θα πρέπει να παραμείνει το θέμα ανοιχτό πέρα τώρα από το αν είμαστε εμεί αρμόδιοι, όχι μάλλον ε, αν ε, έχει να κάνει με το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε βάθο. Ε, και όπω το είπαμε στην αρχή, είχαμε προσκαλέσει του συναδέλφου τη Επιτροπή Μεταφορών να συμμετάσχουν στι εργασίε μα, αλλά ακριβώ είχαν τη συνάντηση τη δική του ταυτόχρονα. Γι' αυτό ακριβώ δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν εδώ απόψε στη συνεδρίασή μα. Γίνεται δεκτή η πρόταση Μποστινάρου η έκθεση για γνωμοδότηση να πάει και στην Επιτροπή Μεταφορών. Προς στιγμή να διακόψουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες, να μην δούμε ποιος άλλος είναι αρμόδιος, να δούμε τη δικιά τους γνωμοδότηση της επιτροπή Μεταφορών και μετά θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε εμείς. Αυτά, σας ευχαριστώ. Συγγνώμη και πάλι για την καθυστέρηση με την οποία ξεκινήσαμε να εξετάζουμε τις, ε, την αναφορά σας και ελπίζουμε όμως ότι θα ξεκινήσουμε έτσι και θα μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση στα θέματα τα οποία θίξατε. Αυτά και σας ευχαριστούμε.